και την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Μας έχει ετοιμάσει και ένα φυλάδιο όσα θα το βρείτε και τυπωμένο στην αίθουσα αλλά και στους φακέλους της συνεδρίασης. Κύριε Γκουρία, καλώς ήρθατε, με χαρά σας υποδεχόμαστε. Uh, uh, yeah, better. Um, thank you, Mr. Chairman. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ξανά μαζί σας. Δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα. Είναι η τέταρτη, πέντε φορά, πέμπτη φορά. Είναι πάντως πάρα πολύ καλό που είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη φορά όμως παρακαλώ να ξεκινήσουμε λίγο αργότερα, να με καλέσετε λίγο πιο αργά. Εν πάση περιπτώσει, ε, η οικονομική επιθεώρηση ε, της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Κάναμε δύο ξεχωριστές επιθεωρήσεις. Μερικές φορές φαίνεται λίγο τεχνητό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αποτελεί αίτημα της ιδίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενεργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν υπάρχουν ε, διαθέσιμα τα δύο έγγραφα ε, και όπως ε, καταλαβαίνετε επί της ουσίας δεν παρουσιάζουν πολύ μεγάλες διαφορές μετά από πολλά χρόνια κρίσης η οικονομική οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, έχουν μειώσει την ενεργεία στο 7,1% που βρίσκονται δηλαδή σε επίπεδα προκρίσης. Ε, ε βεβαίως θέλουμε οικονομικό, έχουμε οικονομικό στόχο της τάξης του 2% και για φέτος και για του χρόνου. Η οικονομική ανάκαμψη έχει ενισχύσει τις οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο τρίτα των Ευρωπαίων, σύμφωνα με το Ευρωμαρόμετρο του προηγούμενου Απριλίου, θεωρούν ότι οι χώρες τους έχουν ευεργετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ε, σε 35 ε, χρόνια είναι το υψηλότερο ποσοστό και επομένως αυτό είναι πολύ καλό, είναι καλό νέο, αποτελεί ε, υποστήριξη του κόσμου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχουν, έχουν, υπάρχει βεβαίως μια ανισομερή κατανομή όσον αφορά τις ευάλωτες περιοχές και υπάρχουν κάποιες περιφέρειες της Ευρώπης οι οποίες έχουν ακόμα υψηλή ανεργία και ε, οικονομική ε, αδυναμία και σε ορισμένες ε, χώρες παρουσιάζεται αύξηση της δύναμης των αντιευρωπαϊκών κομμάτων και βεβαίως διαβάζοντας και τα νέα στις εφημερίδες το καταλαβαίνουμε αυτό. Ε, όσον αφορά την αναχώρα, τις αναχώρα επιθεωρήσεις, ε, πρέπει να πούμε ότι ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να θωρακιστεί καλύτερα η Ευρωζώνη όσον αφορά μελλοντικές, μελλοντικούς κλειδονισμούς και κρίσεις και βεβαίως αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο εδώ είναι ας πούμε η ενσωμάτωση, η ολοκλήρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ε, τραπεζικών ε, προϊόντων κλπ. Περισσότερη Ευρώπη, καλύτερη Ευρώπη, ε, την στιγμή που διεθνώς οι πολυμερείς σχέσεις υφίστανται πίεση. Ακριβώς αυτή η πολυμέρεια μας ενδιαφέρει και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Θα ήθελα τώρα να σας αναφέρω ορισμένα από τα κύρια μηνύματα. Πρώτα απ' όλα η ενδυνάμωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης του, της Ευρωζώνης που αντίθετα από πολλέ προβλέψει. Ε, συνέχισε να λειτουργεί καλά. Βεβαίω παραμένουν ανισορροπίες ε, και ε, η πρόθεση προ την, προς την ολοκληρωμένη νομισματική οικονομική ένωση δεν ήταν ίση και ήδη για όλους. Η Τραπεζική Ένωση επίση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει επιβεβαιωθεί πολλέ φορέ αδιαστόματο Ευρωπαίων ηγετών, αλλά υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο δράση. Ε, και ε, επικεντρώνομαι σε τρεις ε, κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα ενοποιημένη φορολογική βάση έτσι ώστε να μπορέσει να θωρακιστεί η Ευρώπη όσο γίνεται καλύτερα για επόμενες κρίσεις. Τώρα μέσω κάποιου ταμείου, ναι, είναι, θα ήταν μια λογική πρόταση, αλλά βεβαίως το σημαντικό δεν είναι τι όνομα δίνεις σε, σε κάποια λειτουργία, αλλά πώς λειτουργεί ο μηχανισμός αυτό είναι το σημαντικό. Ε, βεβαίως ε, ε, ίσως, ε, τι να σας πω, αν μιλήσουμε για Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, να βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά αυτό δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι τα δύο να είναι συνορματικά και να ενισχύουν ακόμα περισσότερο. Επίσης, το, θα πρέπει να καθοριστεί ένα πρόγραμμα προστασίας καταθέσεων, έτσι ώστε να προστατευτεί πραγματικά η Ευρωζώνη και τρίτον, ένα safe asset ευρωπαϊκού επίπεδου θα πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε ε, να σταματήσει αυτή η αρνητική ανάδραση ανάμεσα στις τράπεζες και τα κράτη. Η Τραπεζική Ένωση βεβαίως από μόνη της δεν αρκεί ε, μακροοικονομικές πιο αποτελεσματικές ε, πολιτικές οι οποίες θα βελτιώσουν πραγματικά τη λειτουργία της Ευρωζώνης απαιτούνται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βοήθησε στη σταθεροποίηση του ευρώ. Αυτή η φράση whatever it takes, ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε, είναι περίφημη πλέον, αλλά και από μόνη της δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ούτε και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στι νέε απαιτήσει του, του τραπεζικού περιβάλλοντος. Νέες φορολογικέ πολιτικές οι οποίε ε, ακόμα ε, δυσκολεύονται και παρεμποδίζονται από υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν υψηλό δημόσιο χρέος αλλά ε, και μηδενικές, μηδενικά επιτόκια. Αλλά αυτό που παρεμβαίνει ανάμεσα στα μηδενικά επιτόκια και την, τις υπόλοιπες καταστάσεις είναι ότι τα νοικοκυριά δεν έχουν καταφέρει ακόμα, ο απλός δεν έχει καταφέρει ακόμα να χρησιμοποιήσει ε, το ευεργέτημα, αν θέλετε, που απορρέει από την κατάσταση αυτή έτσι ώστε ε, να βελτιωθεί και η ίδια η ζωή τους και ε, έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο του ΑΕΠ. Αλλά ξέρετε ότι και πολλές φορές υπάρχει μεγάλη τροτότητα η οποία ούτως ή άλλως δημιουργεί πρόβλημα ακόμα και αν το ΑΕΠ γενικά είναι καλό η επιθεώρηση ε, ε, προτείνει κάποιες ε, προτάσεις όσον αφορά την ανεργία, όσον αφορά ένα ταμείο επανασφάλισης, επίσης και συγκεκριμένες μεταφορές προς ορισμένες χώρες. Οι πρόσφατες προτάσεις της Κομισιόν όσον αφορά επενδυτικές και σταθεροποιητικές δραστηριότητες να, μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον βήμα. Δηλαδή, οι επενδύσεις ε, είναι ε, πολύ καλό ε, πρώτο βήμα και το, το, θέμα και το πρόγραμμα της επανασφάλισης και αυτό είναι ένα δεύτερο καλό βήμα. Επίσης, απλούστευση των φορολογικών κανόνων ε, μέσα από έναν πιο απλουστευμένο κανόνα που θα ε, δίνει ε, δυνατότητα σύνδεσης με το χρέος. Επίσης, εμείς πιστεύουμε ότι στα πλαίσια της πολιτικής θα πρέπει να έχουμε περισσότερο καρότο και λιγότερο μαστίγιο, αν μου επιτρέπετε την παρομοίωση. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, τώρα τα ε, ε, corporate bonds είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερα από τον, τα, τα δάνεια τα τραπεζικά στους διαφόρους ομίλους. Στην Ευρώπη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υποχρησιμοποίηση των corporate bonds και ε, για να αναπτυχθεί ε, και για να αναπτύξουμε την αγορά μας στην Ευρώπη παραδοσιακά ε, βασιζόμαστε περισσότερο στην τράπεζα και στην εργασία των τραπεζών και εδώ πρέπει να γίνει δουλειά για να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Η παραγωγικότητα, πώς, πόσες φορές να σας το πω, παραγωγικότητα και ξανά παραγωγικότητα και ξανά μανα ε, ένας ε, άλλος ε, παράγοντας λοιπόν είναι της ελλειπούς παραγωγικότητας που οδηγεί σε χαμηλά στάνταρ επίπεδα ζωής. Ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να αρθούν εμπόδια ε, σε συγκεκριμένους κεντρικούς τομείς έτσι ώστε οι ανταλλαγές να είναι πιο εύκολες. Ε, θα πρέπει, και το αναφέρουμε αυτό και στην επιθεώρηση, θα πρέπει οι υπηρεσίες να είναι εύκολες. Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 75% στις χώρες μας, της οικονομίας των χωρών μας και εμείς συνέχεια δημιουργούμε προβλήματα, δημιουργούμε δημιουργούμε προβλήματα με τα πετρέλαια, δημιουργούμε προβλήματα με τη μεταποιητική βιομηχανία. 75% της οικονομίας ε, ε, αντιπροσωπεύεται από τις ε, υπηρεσίες, επομένως πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό. Το θέμα των υπηρεσιών λοιπόν είναι θεμελιώδου σημασίας και εδώ ακόμα στον τομέα αυτό υπάρχουν πάρα πολλές ε, ε, ε, πάρα πολλοί περιορισμοί. Επίσης, ενέργεια, στην ενέργεια, στον ηλεκτρισμό, στις τηλεπικοινωνίες, ακόμα βασιζόμαστε σε εθνικούς κανόνες αντί να έχουμε μια γενικότερη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Η ψηφιοποίηση, πολύ σημαντικό θέμα και διασυνδέεται και με την παραγωγικότητα. Πριν από λίγο έβλεπα ότι στη δεκαετία του 90 Μέχρι και το 2007 η παραγωγικότητα ήταν πάνω από 2%. Το 2007 μέχρι το 2017 η παραγωγικότητα, ε, η αύξηση παραγωγικότητα ήταν κάτω από 1%, δηλαδή από πάνω από 2% έφτασε σε κάτω από 1%. Ε, και ε, στην Ευρωζώνη έχουμε φτάσει στο 0,4%. Καταλαβαίνετε, ε, ε, αυτό νομίζω δείχνει το πρόβλημα της μείωσης της αύξησης παραγωγικότητας, αλλά με αυτά τα ποσοστά δεν είναι πλέον βιώσιμη η αύξηση παραγωγικότητας και επομένως μπορεί κανείς να έχει ανάπτυξη βάσει κάποιων σεναρίων, αλλά ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια και η επενδύσεις επενδύσεις έχουν ε, ε, μείνει πίσω και η παραγωγικότητα επομένως έχει μείνει πίσω και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για την μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξη. Η ψηφιοποίηση έλεγα ε, οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. 40% των ενηλίκων ακόμα δεν έχουν ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες και βεβαίως θα πρέπει να δημιουργηθεί και η απαραίτητη υποδομή ακόμα, η οποία ακόμα είναι ελλειπής. Θα πρέπει επίσης ε, στην Ευρώπη να αναπτυχθούν ε, τα εργαλεία τα οποία θα παρακολουθούν ε, τις ψηφιακές και άλλες δεξιότητες. Θα πρέπει να υποβοηθηθεί ο κόσμος έτσι ώστε να αποκτήσει αυτές τις ψηφιακές και άλλες δεξιότητες. Αλλά χρειάζεται και η υποδομή. Προϋπολογισμός τώρα. Ε, οι μεταρρυθμίσεις του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να οδηγήσουν σε ε, γρηγορότερη και πιο συμπεριληπτική ανάπτυξη. Ε, εμείς πάντα υπογραμμίσαμε ότι υπάρχουν και κάποιες νέες ανάγκες. Μάλιστα, εδώ έχουμε σε αυτό το έγγραφο που σας δείχνω και ένα γράφημα το οποίο δείχνει ότι σε πραγματικό αριθμούς και λαμβάνοντα υπόψη το μέγεθο τη Ευρωπαϊκή οικονομία, ο προπολογισμό διαρκώ ε, ε, μειώνεται. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν ζητάει υψηλότερου αριθμού, αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι ε, και λόγω του Brexit η ανάγκη μεταρρύθμισης είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ε, ίσως μετά το, 20, μετά το 2020 θα πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί αυτό το μεγάλο κενό που θα δημιουργηθεί. Ε, όσο έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για, την, για τον νέο προϋπολογισμό και επομένως είναι η κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε να ξανασκεφτούμε την αναθεώρηση. Επίσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον προπολογισμό η δυνατότητα ε, ε, των χωρών να πληρώσουν. Οι πόροι θα πρέπει επίσης ε, να αναζητηθούν σε πλαίσια, στα πλαίσια της ε, της πολιτικής συνοχής ε, και της ε, ΚΑΠ θα πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξισορρόπηση των διαφόρων περιοχών, περιφερειών της Ευρώπης. Η έρευνα και ανάπτυξη αυτή τη στιγμή αποτελεί το 14% του προϋπολογισμού αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί έτσι ώστε να αυξηθεί και το δυναμικό. Ο ευρωπαϊκός προπολογισμός θα πρέπει να κάνει περισσότερα από αυτούς που έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τις τεχνολογικές εξέλιξεις και την καινοτομία. Επί παραδείγματι, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να προσφέρει βοήθεια στους εργαζομένους και να διευρυνθεί το πεδίο του έτσι ώστε να καλύπτει και εκείνους τους οποίους ε, απειλεί η αυτοματοποίηση. Οι περιφερειακές επίσης διαφορές σε ΑΕΠ κατά κεφαλήν είχαν τάση μειωτική μέχρι την κρίση. Από την κρίση και μετά έχουν διευρυνθεί και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όπου εμφανίζεται κρίση, αμέσως ανοίγει η ψαλίδα των ανισοτήτων. Εδώ όμως είχαμε τη μητέρα όλων των κρίσεων. Έχουν περάσει 10 χρόνια και ακόμα έχουμε ορατά, ορατές τις συνέπειες της κρίσεως και γι' αυτό ανοίγουν ακόμη περισσότερο οι διαφορές, οι ανισότητες και σε περιφερειακούς όρους και όχι μόνο σε όρους ε, σύγκρισης μεταξύ κρατών αλλά και στο εισόδημα και στον πλούτο αλλά και στην περιφερειακή ανάπτυξη και μεγαλύτερες διαφορές και ανισότητες. Ένα τρίτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πηγαίνει στην περιφερειακή πολιτική. Τεράστιο ποσό. Ένα τρίτο ή ουδήποτε ποσού ή προϋπολογισμού, οπωσδήποτε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μικρό, λέει ο κύριο Γκουαλτιέρο, ο προπολογισμό. Ναι, όντω είναι μικρό ο προπολογισμό. σω θα πρέπει να έχετε και μεγαλύτερο, λέει ο κύριο Γκουρία. Αλλά δεν είναι θέμα μόνο ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Είναι θέμα ευ εθνικής Δηλαδή πρέπει να αποδοθεί αυτό το 1 τρίτο σε μακροπρόθεσμα σχέδια όπω είναι η εκπαίδευση, οι υποδομέ, οι επενδύσει. Έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί εξίσωση του επίπεδου ε, και βέβαια πρέπει να εξεταστεί όχι μόνο το μέγεθος αλλά και το πώς δαπανώνται τα ποσά αυτά. Εκεί θα κρυθεί η ποιότητα. Με έργα καλά που έχουν ικανοποιητική συγχρηματοδότηση μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη απίκηση. Και έτσι κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάντα ένα εγχείρημα εν εξελίξη. Θα έλεγα είναι ένα διαρκές εργοτάξιο. Μία σκαλωσιά Εσαφοντάζ στα γαλλικά έτσι δεν είναι. Σκαλωσιά. Ξέρετε ότι είμαι Μεξικανός. Στο Μεξικό λέμε «Α, χρήματα πολλά, Ευρώπη, να πάμε η μέση τάξη, να πάει ταξίδι 14 μέρες». Θα πάμε σε 21 πόλεις. Μέσα σε 14 μέρες θα δούμε 21 πόλεις. Έτσι έβλεπε η, μέση αστική τάξη την, ε, ένα ταξίδι προς την Ευρώπη. Και μετά πάει κανείς και βλέπει την Ότροντάμ την Παναγία των Παρισίων, τον τόμο του Μιλάνου, τον καθεδρικό της κολονίας. Μέσα σε, ε, ε, μέσα σε ένα περίβλημα από σκαλοσιές βλέπουμε τον καθεδρικό αυτόν, μέσα στη σκόνη, με τα μηχανήματα που τρίβουν συνέχεια και λέει ο επισκέπτης από τόσο χρόνο ετοίμαζα να πάω και δεν μπορώ να δω τα, ε, έργα τέχνη τα γλυπτά και τα λοιπά και είναι καλυμμένα και μετά ξανάρχεται τρία χρόνια μετά και λέει «Α, τώρα που έχουν αποκαλυφθεί, τι έργο τέχνης είναι αυτό, τι αριστούργημα είναι αυτό». Γιατί τους Ευρωπαίου μπορεί κανεί να του κατηγορήσει για οτιδήποτε, αλλά όχι ότι κάνουν πράγματα βιαστικά ή γρήγορα. Μπορεί να αργούν, αλλά όταν τα κάνουν, τα κάνουν εξαιρετικά. Και εγώ λέω πάντα η Ευρώπη ξανά σχεδιάζεται, ξανά διαμορφώνει τον, ε, το εσωτερικό της, τον εαυτό της, τα θεσμικά της όργανα. Αλλά βεβαίως βιαστικά δεν, γρήγορα δεν προχωρεί. Και εδώ ακριβώς έχουμε το ζήτημα, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αξιολογήσουμε τη διαδικασία της ενοποίησης. Είναι διαρκής προσπάθεια, διόρθωση ξανά, διόρθωση. Δεν φταίει η σκαλωσιά. Οπωσδήποτε δεν προχωράει γρήγορα αυτό το εγχείρημα, αυτό το εργοτάξιο, αλλά γεννά κάτι το καταπληκτικό, το μοναδικό, το υπέροχης αξίας, κάτι το οποίο εμπνέει ολόκληρο τον κόσμο. Και άρα περισσότερη Ευρώπη πρέπει να ζητάμε. Περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, στηριχθείτε στην υποστήριξή μας. Στην υποστήριξη του ΩΣΑ για περισσότερη Ευρώπη, και βέβαια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά και τις χώρες της Ευρώπης θέλουμε να βοηθήσουμε, ώστε να φέρουν σε απτούς όρους να υλοποιήσουν αυτό το υπέροχο εγχείρημα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκουρία για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα λεγόμενά σας και πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα και τα πορίσματα της έρευνας που έχει διεξάγει ο ΩΣΑ. Ήσασταν πολύ πιστικός Και δεν είναι εύκολες ε, οι πολιτικές εποχές που διανύουμε και σε αυτές τις δύσκολες πολιτικά εποχές είναι πολύ θετικό να μας λέτε ότι η Ευρώπη ε, θεωρείται από τους έξωθεν παρατηρητές ως υπόδειγμα. Πράγματι, οι σκαλωσιές μας είναι περίτεχνες και χρειάζεται χρόνος για να στηθούν. Η σκαλωσιά για την ε, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες και τους μήνες να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο πράγματι προς την κατεύθυνση που αναφέρατε. Όλοι αυτοί οι τομείς είναι τομείς προτεραιότητα για εμά, για τους Ευρωπαίους. Συμμερίζομαι απολύτω την ανάλυση σα και ελπίζω ότι θα είναι σε θέση ο ΩΣΑ να προσφέρει λύσεις, αλλά και εμείς ως Ευρώπη να προσφέρουμε λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τέσσερα λεπτά θα έχει στη διάθεσή του ο καθομιλητής. Ο κύριος Νίντερ Μάγερ, παρακαλώ. Πολύ δύσκολο σε τέσσερα λεπτά, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα ήθελα να σας ζητήσω ε, κάποιες συμβουλές για την πολιτική από πλευρά όσα για την εμπορική πολιτική και τις εμπορικές συμφωνίες και τις αντισταθμίσεις. Όλα αυτά από τη μία ευνοούν την ε, ευρωπαϊκή οικονομία, από την άλλη μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Πώς θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπονομεύει τις υπεφωνημένες ε, συνθήκες για το διεθνές εμπόριο. Τα αριθμητικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η Αμερικανική κυβέρνηση είναι αντιπροσωπευτικά. Κάποιοι πιστεύουν όχι. Μιλώ για τη θετική επιρροή της ψηφιακής οικονομίας στην οικονομία των ΗΠΑ, η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας εισαγωγών ε, σε σχέση με την προστιθέμενη αξία. Ποια είναι η αποψή σας, ισχύουν αυτά. Και η αλλαγή πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες υπονομεύει τη σταθερότητα της, της ε, οικονομικής πολιτικής ε, σε χώρες που έχουν τεράστια εμπορικά πλεονεάσματα όπως η Κίνα. Αυτά λοιπόν για τα εμπορικά, τα διεθνή εμπορικά. Δεύτερο, για τη φορολογία. Υπάρχει πρόοδος παγκοσμίως στο θέμα αυτό. Οι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει έτσι περαιτέρω. Πώ τη βλέπετε αυτή την προσπάθεια, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Μιλώ για την εφαρμογή του BEPS, του BEP και την ε, πρόταση για τη φορολόγηση σε σχέση με την ψηφιακή οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Κοιτάξτε, ε, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές, λέει ο κύριος Γκουρία. Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις, πράγματι υπάρχουν εμπορικέ εντάσει και όλε αυτέ οι εντάσει και οι ανακοινώσει οι χθεσινέ απειλούν αν όχι να εκτροχιάσουν τουλάχιστον να επιβραδύνουν την ανάκαμψη τη οικονομία παγκοσμίω. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι αυτό τον κίνδυνο, να τον παραδεχόμαστε, να τον αναγνωρίζουμε. Σύσταση λοιπόν του ΟΣΑ είναι η εξή. Προχωρήστε ε, προς το, τις πολυμερείς συμφωνίες. Ακολουθήστε αυτή την οδό. Και θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Το Χάνξαο, το G20, δημιούργησε το Παγκόσμιο Φόρουμ για την ε, ικανότητα υπερβολικού πλεονάσματος σε σχέση με το χάλιβα. Και το λέω γιατί από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Με το χάλιβα, το ατσάλι, το αλουμίνιο, τους δασμούς, θα υπήρχε παρέκκληση, ε, εξαίρεση, δεν θα υπήρχε. 30 μέρες μετά ε, υιοθετήθηκε νέα εξαίρεση. Και τελικά όλα αυτά έγιναν τη στιγμή που διεξαγόταν η Υπουργική Σύνοδος των χωρών του ΟΣΑ. Ε, βγήκε αυτή η ανακοίνωση για την επιβολή δασμών. Ποιε είναι οι επιλογέ μα σήμερα και ποιε ήταν οι επιλογέ μα και τότε που παραμένουν σήμερα για το χάλιβα, το ατσάλι, το αλουμίνιο. Με την εξαίρεση της Κίνας ισχύουν παντού αλλού. Εμείς λοιπόν δημιουργήσαμε αυτό το Παγκόσμιο Φόρουμ. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το Παγκόσμιο Φόρουμ είναι το μέρος, το βήμα όπου θα ασχοληθούμε με την ουσία του θέματος, όχι τις εκδηλώσεις του ζητήματος ή του προβλήματος. Οι εκδηλώσεις του προβλήματος είναι ότι υπάρχει υπερβολική παραγωγή χάλιβα, το 1 τρίτο είναι πλέον ασματική σε τόνους 2,4 εκατομμύρια πλεονάζουσα παραγωγή και άρα περίπου το 1 τρίτο πλεονάζει. Γιατί έχουμε υπερδυναμικότητα, υπερπαραδυνατότητα παραγωγής κατά 1 τρίτο, διότι πριν από 10 χρόνια θεωρήθηκε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του 12% ετησίως της Κίνας ή του 3 ή 2% ετησίως της Ευρώπης θα συνεχιζόταν. Και άπαξ και ξεκινήσει αυτός ο τροχός δύσκολα σταματάει. Και μετά σε πολλά μέρη και ειδικά στην Κίνα δεν έχουμε τα επόμενα σημάδια για να προχωρήσει η οικονομία και η αγορά στην επόμενη φάση, αλλά ανθεί συνεχώς και αποκλειστικά και μόνο ο κατασκευαστικός τομέας. Άρα η ουσία του ζητήματος είναι πώς θα αντιμετωπίσει κανείς την πλεονάζουσα παραγωγή. Ε, οι εκδηλώσεις του προβλήματος είναι ότι επιβάλλονται δασμοί. Αυτό είναι παρεπόμενο, παρενέργεια αν θέλετε. Και ένας δασμός μετά από τον ένα φέρνει άλλο δασμό από τον άλλον και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι η πλεονάζουσα παραγωγή. Προχθές με ενημέρωσαν ότι οι πρόεδροι του, του G20 της φετινής χρονιάς, δηλαδή η Αργεντινή, αποφάσισε να αναβάλει τη σύνοδο σε επίπεδο που θα είχαμε την επόμενη εβδομάδα στο Παρίσι για το θέμα του Χάλιβα. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιοι από τους βασικούς παίκτες επιβάλλουν δασμούς ο ένας τον άλλον και απειλούν να επιβάλλουν και άλλους δασμούς, δυο και τρεις φορές υψηλότερους και αυξημένους και ως εκ τούτου αυτή η ατμόσφαιρα δεν είναι εξαιρετικά επικοδομητική για να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια λύση, υπάρχει ένα θεσμικό όργανο, πολυμερές θεσμικό όργανο που συστήθηκε από το G20, στο οποίο μετέχει η Κίνα και η ΙΠΑ. Το δημιουργήσαμε αυτό στη σύνοδο G20 στο Hangzhou στην Κίνα και μετά πήγαμε στο Αμβούργο πέρσι και επικυρώσαμε τη δημιουργία του ε, οργάνου αυτού. Γιατί μέρος της δήλωσης των ηγετών ήταν ότι θα πρέπει να συζητούμε στο πλαίσιο του Global Forum, του Παγκόσμιου Φόρουμ για την πλεονάζουσα ε, δυνατότητα παραγωγής ε, του χάλιβα. Και μετά κάποιοι επέβαλαν δασμούς αντί να έρθουν και να τα συζητήσουν αυτά στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Φόρουμ. Άρα η συμβολή μας είναι ακολουθήστε την πολυμερή άγουσα, είναι ο μόνος τρόπος να λυθούν τα ζητήματα. Πώς λύνει κανείς εμπορικά ζητήματα τα οποία εξορισμού είναι πολυμερή, πώς λύνει επενδυτικά ζητήματα που εξορισμού είναι πολυμερή, πώς λύνει μεταναστευτικά προβλήματα που εξορισμού είναι πολυμερή, πώς λύνει κλιματολογικά θέματα που το κλίμα και η αλλαγή του δεν γνωρίζει σύνορα. Τα σύνορα είναι ανθρώπινη κατασκευή, ενώ οι εκπομπέ των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου δεν σταματάνε στο σύνορο, το οποίο είναι νοητό. Άρα η απάντηση είναι πολυμέρεια, πολυμερής αντιμετώπιση, τη στιγμή που αυτή η αντιμετώπιση τίθεται ένα αμφιβόλο. Τώρα, για τη φορολογία αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, BEP, κανονισμός και ε, φορολόγηση της ψηφιακής δραστηριότητας. Καταπληκτικά τα αποτελέσματα για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν λάβει 92 εκατομμύρια. Εν θα λάβουν 240 εκατομμύρια χάρη του BEP, δισεκατομμύρια. Όμως δεν υπάρχει συμφωνία σήμερα για τη φορολόγηση της ε, δραστηριότητας στην ψηφιακή οικονομία και θα διατυπώσουμε και θα συντάξουμε την τελική έκθεση ως όσα για το θέμα αυτό μάλλον του χρόνου. Παρόλο που έχουμε χρόνο μέχρι το 2020, μας ασκείται πίεση να δημοσιεύσουμε την έκθεση το 2019 και θα το πράξουμε. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ναι, σας ευχαριστώ. Ε, πρέπει να περιορίζουμε το χρόνο μας για να μπορέσουν και άλλοι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο. Κυρία Μπερές, στα τέσσερα λεπτά παρακαλώ το πολύ πάντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ στα αγγλικά. Λυπάμαι που είστε Μεξικανός, αλλά θα σας προτείναμε επικεφαλής ε, ψηφοδελτίου για τις προσεχείς ευρωεκλογέ. Κάποιο κόμμα θα σας ήθελε οπωσδήποτε. Και τώρα μιλάω στη μητρική μου γλώσσα, εκφράζοντας την ικανοποίησή μου που η Ματίλντ Σαμουρέ, μια από τις δικές μας συνεργάτηδες, θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί μέσα σύντομα. Να τι εκεί είναι. Μα τη βουτήξατε αλλά σας την παραδίδουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και χαρά. Μιλήσατε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ναι, είπατε ότι δεν ε, ε, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Είπατε ότι δεν κρίνεται τίποτα από το όνομα. Βεβαίω, αλλά έχει και αυτό κάποια σημασία. Ε, αν θέλετε, βοηθήστε μα. Με ένα νέο όνομα, ενδεχομένω. Ταμείο Σταθεροποίηση. Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθεροποίηση, για να μην υπάρχουν και να μην υπάρχει και δημιουργική ασάφεια. Και για να επανέλθω στην ερώτηση του κυρίου Νίτερ Μάιερ για το διεθνέ εμπόριο. Εκεί βλέπουμε πως είμαστε σε ένα σημείο καμπής και όχι μόνο επειδή εξελέγει στην Προεδρία των ΗΠΑ ο κύριος Τραμπ, αλλά και γιατί οι πολυμερείς σχέσεις πια έχουν αλλάξει όρους σε σχέση με την εποχή της θέσπισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Έχουμε νέους παράγοντες πολύ πιο ισχυρούς. Έχουμε νέα τεχνολογία που αλλάζει τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, έχουμε δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη Σύνοδο COP21. Και άρα, μία προσέγγιση σε σχέση με το κλίμα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και δεσμεύσεις οι οποίες επηρεάζουν την φύση του εγχειρήματο που επιδιώκουμε. Και γι' αυτό ορισμένοι από εμά μιλούν για μία ε, προσαρμογή σε τέλη άνθρακα, για τα τέλη άνθρακα στα σύνορα. Δηλαδή, μήπως υπάρχει δυνατότητα, το βλέπετε εσείς, αντί να γυρίσουμε στις συνθήκες των ελεύθερων συναλλαγών, στο θέμα των ε, κλιματικών αλλαγών να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Γιατί μπαίνουμε στο κλαμπ, ε, στη λέσχη των ελεύθερων συναλλαγών εφόσον σεβόμαστε τους κανόνες και γιατί είμαστε προσιλωμένοι στις ε, αρχές ε, των ελεύθερων συναλλαγών αλλά μήπως θα έπρεπε πέραν της λέσχης των ελεύθερων συναλλαγών να φτιάξουμε και μια λέσχη κλιματικής αλλαγής όπου αναπτύσσουμε περισσότερο τους πολυμερείς κανόνες με βάση βέβαια και τις ιδέες του Λιονέλ Φοντανή που όμως θα πρέπει παράλληλα και να αναπτυχθούν περισσότερο καθώς επιλύουν ή επιτρέπουν την επίλυση ζητημάτων όπως αυτό του χάλιβα που και εσείς επισημάνατε. Ο κύριος Γκουρία. Έχουμε ήδη ε, συμφωνία του Παρισιού για τη μείωση εκπομπών και έχουμε ήδη επίγνωση ισχυρή μάλιστα ε, επίγνωση ότι πρέπει να ε, έχουμε οικολογική συνείδηση και άλλωστε έχουμε ισχυρή οικολογική πράσινη συνείδηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι ότι πέρα από την ανακοίνωση ε, των Αμερικανών ότι θα φύγουν από τις συμφωνίες COP, διαπιστώσαμε ότι εντός των Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε μια σημαντική επιστροφή και μάλιστα δυναμική των αρχών των πολιτιών και των πόλεων Μάλιστα στο, το Σεπτέμβριο στην Καλιφόρνια θα έχουμε μια μεγάλη συνάντηση όλων των δημάρχων. Έχουμε επίση και τον ιδιωτικό τομέα, γιατί εν τέλει ο ιδιωτικό τομέα είναι αυτό, ο οποίο θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου τη μείωσης των εκπομπών. Νομίζω λοιπόν ότι το γενικότερο περιβάλλον είναι πολύ θετικό, αλλά βεβαίω το μεγάλο ερώτημα είναι το εξή pour euh, Πώς να σας το πω. Καταλαβαίνουμε, διαστανόμαστε τον επίγοντα χαρακτήρα. Αυτό νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο την αίσθηση του επίγοντος χαρακτήρα. Ε, ναι, υπάρχουν νέοι πρωταγωνιστές, ναι, υπάρχουν μερικοί εξ αυτών που είναι πολύ δυνατοί, ε, όμως πιστεύω ότι σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πολλά ε, στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι ο άνθρακας θα πρέπει να ε, κοστίζει πολύ. Αυτό είναι μεγάλη αποτυχία. Ε, για την ώρα δεν έχουμε υψηλή τιμή για τον άνθρακα. Έχουμε μονάχα κάποιους μηχανισμούς τύπου ανταλλαγής εκπομπών, ETS ε κτλ. Αλλά οι τιμές του ε, ε, άνθρακα είναι ακόμα πάρα πολύ χαμηλές και έτσι, και έτσι δεν αναπτύσσονται κάποιες εναλλακτικές. Ο κύριος Σάπλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είναι, ε, λέει ο κύριος Κλίντσε, πολύ ε, ενθαρρυντικά ένας Μεξικανός να μιλάει με τόσο ενθαρρυντικά λόγια και τόσο αισιόδοξα λόγια για την Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά έχω και κάποιες ερωτήσεις. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι δύο τρίτα των πολιτών πιστεύουν στην Ευρώπη και υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή ιδέα, αλλά στην πραγματικότητα όλο και περισσότεροι ψηφίζουν για ευρωσκεπτιστικά ε, ε, κόμματα, με τελευταίο παράδειγμα ε, την Ιταλία. Δεύτερο σημείο όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι ήδη πόροι, αλλά αυτοί οι ήδη πόροι από πού θα πρέπει να προκύπτουν. Τρίτον, υποφέρουμε από μεγάλη ζημία ε, λόγω εγκληματικών δράσεων. Χάνουμε κάθε χρόνο περισσότερο από 50 δις ε, ευρώ λόγω της ε, διευρυμένης απάτης. Η Ευρώπη χάνει πάρα πολλά χρήματα πλέον λόγω εγκληματικών δράσεων όσον αφορά την χρήση κρυπτονομισμάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα στην ουσία να συγκρατήσουμε τις απώλειες αυτές ή να τις αποτρέψουμε, πώς μπορούμε να ζητήσουμε από τους ε, ε, πολίτες να δώσουν περισσότερα για τον κοινό προπολογισμό. Τελευταίο σημείο. Αναφερθήκατε στην ιδέα της ε, Κομισιόν για την εισαγωγή αυτών των συστημάτων ε, ε, ε, διασφάλισης καταθέσεων κλπ. Δεν νομίζετε ότι αυτά τα save assets θα έπρεπε να τα είχαν, αυτά που ονομάζονται save assets, θα έπρεπε ήδη οι τράπεζες οι ίδιες να τα έχουν υλοποιήσει, γιατί εδώ θυμάμαι και τις διάφορες διασφαλίσεις για, για τα ενυπόθηκα δάνεια που υπήρχαν στις ΗΠΑ και είδαμε που καταλήξαμε απάντηση. Ναι, γι' αυτό φαίνεται ότι εγώ μιλάω συνέχεια, γιατί μετράνε την ερώτησή σας και μετά δεν σταματάει το χρονόμετρο. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι είμαι Μεξικανός ε, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι, ε, δεν έχω αλλοιωμένη αντικειμενικότητα. Είμαι πολλά χρόνια επικεφαλής του ΩΣΑ και έχω δει τις εξελίξεις. Θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Όταν ήμουν 18 χρονών, πολλά χρόνια πριν, 50 χρόνια πριν συγκεκριμένα. 50 χρόνια πριν. Ήμουνα 18 χρονών λοιπόν και μετέφραζα μία μπροσούρα, ένα φυλάδιο της Ομοσπονδιακής ε, Ηλεκτρικής Εταιρείας ε, του Μεξικού ε, που, θα, είχε σκοπό να βγάλει κάποια ομόλογα σε ΕΚΙΟΥ, σε Ευρωπαϊκές Λογιστικές Μονάδες. Πόσα χρόνια πριν, φανταστείτε, ήμουν εγώ ακόμα μικρό παιδί. Επομένως εγώ στη ζωή μου και στη διάρκεια της ε, ζωής μου έχω ε, έχω ε, καταγράψει τις προσπάθειες της Ευρώπης να έχει τέτοιου είδους λογιστικές, ας νομισματικές μονάδες. Ήταν οι ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες πριν και από το ΕΚΙΟ ακόμα. Επομένως, ο σχηματισμός ε, της ε, Ευρώπης ε, είναι ακόμα εν Και εγώ, και εγώ έχω παρακολουθήσει λοιπόν αυτό το γίγνεσθε της ευρωπαϊκής πραγματικότητας από όταν ήμουν παιδί. Το Ευρωμαρόμετρο λοιπόν λέει ότι δύο τρίτα υποστηρίζουν την Ευρώπη. Τώρα τι ψηφίζουν είναι διαφορετικό. Ναι, αλλά ξέρετε, αυτό το θέμα των εκλογών και το, το, του αποτέλεσμα των εκλογών προκύπτει λόγω της ιοπηρή πλειοψηφίας που δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί χάσαμε τον Brexit, μα γιατί 60% των νεαρών, των νέων ανθρώπων δεν μετακινήθηκαν καν, δεν θεώρησαν απαραίτητο να πάνε να, ψηφίσουμε, να ψηφίσουν. Ε, άρα δεν χάνουμε τη μάχη μονάχα λόγω της έλλειψης ε, εμπιστοσύνης ε, στους θεσμούς της Ευρώπης, ε, αλλά χάνουμε την, ε, την μάχη της εμπιστοσύνης ε, στην δημοκρατία. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αν πάνε να ψηφίσουν θα ψηφίσουν κατά, είναι ότι δεν πάνε καν να ψηφίσουν. Επομένως θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος και εμείς θα πρέπει καλύτερα να το κοινωνήσουμε προς τον κόσμο ότι ε, ε, τα διακυβεύματα είναι μεγάλα. Το, το κύριο διακύβευμα, αυτό που παίζεται στην ουσία είναι το μέλλον μας, είναι η ζωή μας. Και ακριβώς αυτό το μέλλον, αυτή η ζωή απειλείται από τις ε, ακραίες θέσεις Ε, και είδαμε τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία, το, αυτό το μη αναμενόμενο ε, αποτέλεσμα εκλογικό στην Ιταλία, τα όσα συνέβησαν τα, πολιτικά πράγματα και τα εκτενόμενα στην Ισπανία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ε, ένα μαλέζ, μία άσχημη κατάσταση. Τα κρυφονομίσματα, κρυπτονομίσματα δεν είναι νομίσματα, είναι ενεργητικό, είναι assets και ως τέτοια μπορούν να ε, πολλούνται και να αγοράζονται. Πρέπει όμως να προστατέψουμε τους επενδυτές γιατί αυτά δεν είναι νομίσματα. 50 εκατομμύρια ε, απάτη ΦΠΑ. Ναι, αυτό είναι εγκληματική πράξη. Αλλά ακριβώς γι' αυτό ε, λέμε ότι υπάρχει το ζήτημα ε, της ε, φορολογίας, σωστή, σωστό φορολογικό μίξ και ε, όσον αφορά τώρα τις, ε, τους ε, τίτλους ασφάλειας, δεν, είναι, δεν συμφωνώ μαζί σας. Το ενυπόθηκο δάνειο, ε, στα ενυπόθηκα δάνεια είχαμε προβλήματα λόγω της ίδιας της κατάστασης. Εδώ μιλάμε όμως για ομόλογα διαφορετικού είδους. Υπάρχουν στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, αλλά το, το ζήτημα είναι ότι αυτές οι χώρες έχουν ήδη πλεόνασμα, επομένως δεν μετράει. Ευχαριστώ Φίλιπ Λάμπερτς. Είστε πάντοτε ευπρόσδεκτος κύριε Γενική Γραμματέα. Μου αρέσει που μιλάτε με ειλικρίνεια και αυτό είναι καμπανάκι αφύπνισης. Πρώτον, για την ανεργία θέλω να σας ρωτήσω. Μιλήσατε με θετικά λόγια για την εξέλιξη της ανεργίας. Εγώ όμως κοιτάζω τα ποσοστά απασχόλησης και μάλιστα με ε, απασχόλησης πλή, πλήρους απασχόλησης και τα αριθμητικά στοιχεία δεν είναι καθόλου καλά. Το 75% είναι το καλύτερο νούμερο στις καλύτερες χώρες. Στην Ιταλία το 55% έχει μόνιμη απασχόληση από αυτών που εργάζονται. Και αυτό είναι πολύ καλύτερο καλύτερος ε, για το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Η χαμηλή ποιότητα των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται είναι λόγος ανησυχία για εμάς. Ουσιαστικά έχουμε γίνει όλοι και όλες οι νέε ε, δουλειές έχουν γίνει σαν την Uber την εταιρεία ταξί. Ε, δεν υπάρχει υποχρέωση αμοιβή αν δεν παραχθεί κάποιο έργο, ούτε υπάρχει υποχρέωση παραγωγή συγκεκριμένου έργου. συμβόλαια δηλαδή μηδενική αμοιβή οξύνονται οι ανισότητες. Ενώ τελικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τις επενδύσεις και με αυτό το οποίο συνέβη μειώθηκαν οι ανισότητες. Σε λιγότερο δραματικές περιπτώσεις στη Φιλανδία στις αρχές του 1990 υπήρξε κρίση και τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για να αντιμετωπιστεί η κρίση ουσιαστικά οδήγησαν στο να μειωθούν οι ανισότητες και αυτό είναι καλό πράγμα. Δεν είναι δηλαδή ε, ε, κάτι το μοιραίο που μόνο έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι πολιτική επιλογή το ποιος θα πληρώσει την κρίση. Ε, οι πλούσιοι πληρώνουν λιγότερο σήμερα την κρίση και νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά πολιτική επιλογή. Δεν είναι πανάκια, ούτε μονόδρομος. Εκτιμώ ιδιαίτερο τη δουλειά που κάνει ο ΩΣΑ, ειδικά για τον ΠΕΠΣ, για τον BEP. Ε Όμως, έχω την εντύπωση ότι Έχουμε από τη μία την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λειτουργεί ως νομοθέτης και όταν αποφασίσει σε κάποιο τομέα να προχωρήσει περισσότερο από τα πρότυπα του ΟΣΑ, ο ΟΣΑ από το Παρίσι ανθίσταται. Ενώ όσοι θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο από τα κοινώ συμπεφωνηθέντα πρότυπα θα έπρεπε να μπορούν να το κάνουν, γιατί έτσι ασκείται και πίεση στους υπολείπου να κινητοποιηθούν περισσότερο. Ποια είναι η άποψή σας από αυτού. Απάντηση. Δεν ε, ανταγωνιζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπληρώνουμε, λειτουργούμε συμπληρωματικά όσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει και να ευθετήσει οδηγίες που θα έχουν βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα ε, δυσκολέψουν την εφαρμογή των μακροπρόθεσμων λύσεων. Λέμε λοιπόν ότι κατανοούμε ε, τι πολιτικέ δυσκολίε Ο Μπρινό Λεμέρ μα λέει ότι θέλει να προχωρήσει ο καλός υπουργό Οικονομικών και μα λέει πρέπει να φορολογήσετε αυτέ τι εταιρείε και συμφωνώ. Δεν μπορούμε να έχουμε εταιρείε που να μην φορολογούνται πουθενά. Πόσο μάλλον εταιρείε που έχουν ε, κέρδη εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να φορολογούνται όπως και οι υπόλοιπες εταιρείε. με το τρέχοντα φορολογικό συντελεστή στη δικαιοδοσία που ανήκουν. Όμως το πώς θα φορολογηθούν, το πού θα φορολογηθούν, με, το, με ποια βάση, με ποιο συντελεστή φορολογικό, είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο συντονισμού. Ή αλλιώ θα γίνει σαν την αυτόματη ενταλλαγή πληροφοριών και τους φορολογικούς παραδείσους. Αν σε μπλοκάρουν εδώ, θα πας στην άλλη χώρα και μετά στην άλλη χώρα. Αν τελικά όλοι αυτό κάνουν στον κόσμο, τότε δεν θα μπορέσουν να κρυφτούν οι επιχειρήσεις αυτές. Αυτό το κάναμε με τους φορολογικούς παραδείσους και τώρα πρέπει να το κάνουμε με τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Μας πιασκούν πίεση να έχουμε έκθεση το 2019 και όχι το 2020 και θα το κάνουμε για να είναι έτοιμε οι λύσεις. Σήμερα οι Αμερικανοί είναι σε διαφορετική κατάσταση από ό,τι τα παλιά. Θα προτιμούσαν να μας περιμένουν εμά τον ΩΣΑ. Υπάρχει όμω σύγκληση και καλή βούληση. Με την τελευταία φορολογική του μεταρρύθμιση κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση. Οι Βρετανοί προσπαθούν και αυτοί να συμμετάσχουν κάπως είναι στο μετέχμιο. Θέλουν να δουν προς τα πού θα γύρει η πλάστικα ξεκίνησαν με το να θέλουν αυτή τη φορολόγηση, μετά ε, θέλουν να καθυστερήσει. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να ξεκινήσουν για αυτή η δουλειά τη φορολόγηση για την ψηφιακή οικονομία του χρόνου. Εμεί θα έχουμε όμω έτοιμη την έκθεση το 2019 για να καταλήξουμε σε ένα κοινό σύστημα αντιμετώπιση. Ζητούμε από την Ευρώπη να μην κάνει κάτι σε βραχυπρόθεσμη βάση που τελικά θα παρακολύσει και θα αποτελέσει τροχοπέδι τη λύση σε μακροπρόθεσμη βάση. Αυτά για την ψηφιακή οικονομία, για την ανισότητα. Δεν πρόκειται περί πολέμου. Η κρίση ήταν τρομακτική, αλλά ήταν και στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και στο χρηματοπιστωτικό τομέα έχουμε ανθρώπους που είναι σε ευνοϊκή θέση και αυτοί είναι πολύ καλύτερα προστατευμένοι από τους πιο ευάλωτους. Αυτό συμβαίνει στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Όσοι δεν είχαν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα στοιχεία ενεργητικού, τα απαραίτητα ήταν λιγότερο προστατευμένοι. Και άρα η ανισότητα διευρύνθηκε λόγω της κρίσης διότι υπήρχε οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Και ναι, έχετε δίκιο. Μιλούμε για τις πολιτικές, για τους νόμους, αλλά και για το γεγονός ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο έχει αυξήσει το μερίδιο που καταλαμβάνει στο εγχώριο ΑΕΠ κάθε χώρας. Και γι' αυτό ο κόσμος είναι τόσο θυμωμένος και τόσο δυσαρεστημένος. Τώρα για τα ποσοστά απασχόλησης. Διαφωνώ με αυτό που λέτε, ότι ε, έχουμε στην Ιταλία 55% πλήρους απασχόλησης. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Στην Ιταλία είναι ιδιαίτερο χαμηλό αυτό το ποσοστό. Δεν ισχύει όμως παντού. Δεν μπορεί κανείς απαραίτητα να πει ότι μια χώρα είναι σε χειρότερη κατάσταση γιατί η αγορά εργασίας της είναι πιο ευέλικτη. Να σας δώσω το παράδειγμα της Γερμανίας, η οποία έχει εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ατόμων που εργάζονται σε καθεστώς μερική απασχόληση. ιδιαίτερω οι γυναίκε Χρειάζονται οι γυναίκε στη Γερμανία να αυξάνουν το ποσοστό τη πλήρου απασχόλησή του. Ε, πάση περιπτώσει, αυτό δεν σχετίζεται με την ευημερία. Ούτε με την παραγωγικότητα μιας συγκεκριμένη χώρας. Το ότι όταν υπάρχει μεγάλο ποσοστό μερική απασχόλησης δεν υπάρχει ευημερία, γιατί η Γερμανία δείχνει το αντίθετο. Όμως, για το πρόβλημα του κατά πόσο όλα τα επαγγέλματα θα γίνουν σαν την Uber, δεν είναι το θέμα η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, αλλά η προστασία αυτών που εργάζονται σε αυτές τις πλατφόρμες. Δηλαδή, οι απώλειες να είναι υποχρεωτικές για όλους και να διευρύνουμε την προστασία. Ο κύριος Παπαδημούλης, παρακαλώ. ε, κύριε Γενική Γραμματέα, σας καλωσορίζουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω μόνο για ένα θέμα που αφορά στην πατρίδα μου την Ελλάδα πριν λίγες εβδομάδες επισκεφθήκατε την Ελλάδα, είχατε σειρά συναντήσεων, συναντηθήκατε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι προβλέψεις σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, ποια είναι η αποτίμησή σας για τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και κυρίως θα ήθελα να σας ρωτήσω για την ε, ελάφρυση του ελληνικού δημόσιου χρέους όπως έχει συμφωνηθεί στο Eurogroup του Ιουνίου του 2017 και μάλιστα ομόφωνα. Σε δύο ημέρες έχουμε ένα πολύ σημαντικό Eurogroup στις 21 Ιουνίου όσοι εμπλέκονται στο θέμα εκ μέρου των δανειστών προεξοφλούν μια θετική έκβαση και ότι θα είναι το Eurogroup που θα δρομολογήσει την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Θυμάμαι στην Αθήνα τη δήλωσή σας, τώρα πια δεν μιλάμε για Grexit αλλά για exit της Ελλάδας από τα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης. Επειδή ως Μεξικανός και ως Γενικός Γραμματέας του, ΟΗΕ, του, του ΟΟΣΑ, με συγχωρείτε, ξεχωρίζετε για την καθαρή σας γλώσσα, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για την ανάγκη ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους ως κλειδί για την επάνωδο στις αγορές. Ευχαριστώ. Θα έπρεπε να έχουμε προαγάγει ένα μαζικό ένα ε, σχέδιο ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας με μαζική υποστήριξη από την Ευρώπη, τη Γερμανία, τη Γαλλία όταν ήταν 300 δις θα μπορούσε να έχει γίνει μια σημαντική απομείωση για να έχουμε πολύ χαμηλότερο χρέος τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι οι Υπουργοί των Οικονομικών εκείνης της εποχής αποφάσισαν ότι κινδύνευαν οι τράπεζες των δικών τους δικαιοδοσιών και επέλεξαν να προστατεύσουν το τραπεζικό σύστημα που, είχε, που ε, διακρατούσε μεγάλο κομμάτι ελληνικού χρέους για να μην υποστούν τις συνέπειες οι τράπεζες. Άρα τι έκαναν, δάνεισαν στην Ελλάδα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου για να πληρώσει η Ελλάδα, να ξεπληρώσει τελείως το χρέος της προς τους πιστωτές του ιδιωτικού τομέα και μετά αυτό το ιδιωτικό χρέος η Ελλάδα με κάποιες μικρές απομειώσεις το μετέτρεψε βασικά σε δημόσιο χρέος. Το οποίο είναι πολύ πιο ανελαστικό τώρα γιατί δεν μπορεί να γίνει απομείωση από το Δουνουτού, δεν μπορεί να γίνει απομείωση από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και ούτω καθεξής. Άρα ποιο είναι το ζήτημα. Όντως, ναι, η Ελλάδα θα είναι καλύτερα. 2,0 φέτος. 2,3 του χρόνου. Οπωσδήποτε σημαίνει ότι τα πάει καλύτερα. Γιατί χάρη στις μεταρρυθμίσεις της. Γιατί αυτοί οι μεταρρυθμίσεις ήταν πολύ επώδυνες, πολύ δύσκολες και οφείλω να πω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα και ο ελληνικός λαός έμειναν αμετακίνητη σε αυτή την πορεία μεταμορφώνοντας την ελληνική οικονομία σε όρους πιο καλούς, πιο θετικούς, πιο πρακτικούς. Ερώτηση. Χρειάζεται η απομείωση του χρέους. Βεβαίως, ναι, το έχω ξαναπεί. Το λέω κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα, κάθε φορά που μου διατυπώνεται η ερώτηση και το ξαναλέω. Σήμερα είναι δυνατόν να υπάρξει ονομαστική απομείωση του χρέους. Πολιτικά η απάντησή μου είναι σήμερα όχι. Υπάρχουν πραγματικοί παράγοντες που παρεμποδίζουν μια τέτοια εξέλιξη. Η κοινή γνώμη, διεθνής κοινή γνώμη δεν είναι όριμη, γιατί το ζήτημα δεν είναι μία χώρα, αλλά πολλές χώρες που αντιλαμβάνεστε ότι εάν ε, κάποιο έχει περάσει μέσα από μία κρίση, μπορούν να πούνε Α, κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να ταλαιπωρηθούν, να υποφέρουν κτλ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά υπάρχει αυτή η θέση. Τώρα, μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάτι καλύτερο σε όρους τωρινών αξιών, χώρο, περίοδο χάριτος, ε, καθυστέρηση στην αποπληρωμή των, ε, των τόκων, κάτι που θα βοηθήσει την Ελλάδα να ξανασταθεί στα πόδια της, να ανακτήσει την οικονομία της, να προχωρήσει την ανάπτυξη. Ναι, αυτό είναι δυνατόν και αυτό πρέπει να προσπαθήσετε ακόμη να αξιοποιήσετε και να διερευνήσετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Τώρα για λόγους ε, χρόνου θα πρέπει να ακούσουμε ε, περισσότερες ερωτήσεις από περισσότερους συναδέλφους μαζί. Παρακαλώ κύριε Ροζάτη, Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Γενική Γραμματεύ που είστε εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ για την ε, σαφέστατη υποστήριξη προς τις πολυμερείς σχέσεις στο πολυμερές σύστημα. Ιδιαίτερα πολύτιμη αυτή η υποστήριξη, ιδιαίτερα τώρα που υφίσταται τόσες πολλές επιθέσεις. Θα ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις σε σχέση με το δυναμικό απόδοσης και ανάπτυξη ολόκληρο τον κόσμο βεβαίως, αλλά ειδικότερα στην Ευρώπη. Ποιοι είναι οι λόγοι που βλέπετε αυτή τη συγκράτηση στην Ευρώπη ιδιαίτερος, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οφείλεται δηλαδή ε, αυτή η καθυστέρηση στην απουσία επενδύσεων σε δραστηριότητα ε, σε τοπική δραστηριότητα, όπως επισημάνει ο κύριος Λάμπερτς, είναι επιβράδυνση στην ε, παραγωγικότητα. Επίσης, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και στο τμήμα το οποίο στοχεύει στη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Πώς θα μου τον αξιολογήσετε, θεωρείτε, γιατί υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι πρώτα πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση χάρη στην τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων και ότι αν οι χώρες δεν ακολουθούν αυτούς τους κανόνες προφανώς και δεν μπορούν να περιμένουν υποστήριξη γιατί θα έπρεπε καταρχάς να έχουν τηρήσει τους κανόνες και μετά να έχουν την υποστήριξη. Και τρίτον, η δουλειά του ΩΣΑ για την ε, φορολογία. Τι βλέπετε λοιπόν ως ε, ιδανικό ε, λόγο, ιδανική αναλογία μεταξύ άμεσων και έμεσων φόρων, ειδικά δεδομένου ότι οι άμεσοι φόροι όλο και πιο δύσκολα συλλέγονται λόγω της μεγάλης κινητικότητας του κεφαλαίου, της δυνατότητας μεταφοράς κέρδου σε άλλες περιοχές ή χώρες. Πώς βλέπετε λοιπόν τη δυνατότητα της εξασφάλισης των δημοσιονομικών πόρων για τα κράτη, ε, με άμεσους ε, φόρους, με τα άμεση φορολογία ή με έμεση ο κύριος Αρέγγι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκουρία. Εγώ χαίρομαι που σας ε, βλέπω να είστε έτσι τόσο παθιασμένος και τόσο αισιόδοξο, γιατί και τα δύο στοιχεία είναι σημαντικά σε μια τέτοια περίοδο. Εγώ θα ήθελα να ε, κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Πρώτον, ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά την δυνατότητα δημιουργίας προπολογισμού της Ευρωζώνης. Γιατί ενδεχομένως στην διάσκεψη κορυφής της επόμενης εβδομάδας, στο τέλος του μήνα δηλαδή, δεν θα εγκριθούν τρομερά σημαντικά σημαντικά μέτρα αφορά την Οικονομική Νομισματική Ένωση, την, ε, το, Ταμείο Εγγύηση Καταθέσεων κλπ. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν οριμάσει δυστυχώς ε, οι καιροί. Ενδεχομένως όμως ε, υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε στη δημιουργία προπολογισμού για την Ευρωζώνη. Πώς αξιολογείται αυτή τη δυνατότητα. Δεύτερον, λαμβάνοντα υπόψη ότι οι εξαγωγέ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υποφέρουν ε, ως αντίκτυπο αυτών των εμπορικών πολέμων που δυστυχώς υπάρχουν. Ποια ε, σημασία θα είχε η αύξηση των μισθών ως μηχανισμό ενδυνάμωσης της ανάπτυξης. Δεν πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα να έχουμε αύξηση των μισθών έτσι ώστε να προκύψει αύξηση της εσωτερικής ζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Μια τελευταία σύντομη ερώτηση ο κύριο Φραντσούλικα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματεύ, η Ρουμανία ε, είναι η μεγαλύτερη οικονομία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ε, θα ήθελα λοιπόν σύντομα να σας ρωτήσω ποιο είναι το πρόβλημα όσον αφορά ε, την ένταξη της Ρουμανίας στον ΩΣΑ. Προσπαθήσαμε το 4, το 12, το 17. Είναι τεχνικό το πρόβλημα ή μήπως είναι πολιτικό. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα. Η ανάπτυξη βρίσκεται στην, στην παραγωγικότητα, ε, στις επενδύσεις, ε, στις δεξιότητες και το τονίζω, δεξιότητες ε, βεβαίως η αντιμετώπιση της γύρενσης, το θέμα της συμμετοχής των νέων και των γυναικών και όλων, εν πάση περιπτώσει, στην αγορά εργασίας. Και, και ε, ή διαθετικές αλλαγές, ε, γιατί δεν έχουμε πολύ χώρο όσον αφορά τη φορολογική πολιτική, ε, όσον αφορά την διαρθρωτική πολιτική, άρα χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να αυξηθεί το δυναμικό μας. Η, δυνατότητα, η διαδικασία σταθεροποίηση του ευρώ ναι, αλλά βεβαίως θα πρέπει να έχουμε πρόταση για κειμένους κανόνες, οπωσδήποτε και εξορισμού αυτό. Αλλά, αλλά ε, ε, πάντα προκύπτει κάποιο ατύχημα το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στους μηχανισμούς και λέμε όλοι πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και όχι ε, και βεβαίως η κρίση θα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση και θα πρέπει σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις να έχουμε τη δυνατότητα να ε, τις αντιμετωπίσουμε και βεβαίως να έχουμε τη δυνατότητα να αποτρέψουμε τον κίνδυνο στο σύνολο. Τώρα, όσον αφορά την ε, ε, ιδεώδη φορολογική πολιτική. Ε, αυτό δεν υπάρχει, αλλά μπορούμε να μειώσουμε την, της, την επιχειρηματική φορολόγηση, να δημιουργήσουμε δηλαδή περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Αυτή είναι η τάση και ποια είναι η τάση αντιστάθμισης σε περισσότερο ΦΠΑ, περισσότερη επιχειρηματική φορολόγηση, φορολόγηση των εταιριών και και περισσότερες πράσινες ε, ε, ε, φορολογήσεις. Έτσι κινείται ο κόσμος και βεβαίως ξέρουμε ότι και ο τρόπος και η ταχύτητα είναι διαφορετική. Τώρα, στον επόμενο ομιλητή. Οι εξαγωγές δεν υποφέρουν λόγω των εμπορικών πολέμων. Αυτό είναι του χθες η πόλεμη αυτή. Τι να σας πω, ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς πιστεύουμε ότι οι εντάσεις εμπορικές όντως μπορούν να επιβραδύνουν την ανάκαμψη. Αλλά τι να σας πω, αφορούν το 1% της ανάκαμψης. Ε, αλλά αυτό βεβαίως σημαίνει εκατομμύρια ε, άνθρωποι και αφορά την ευζοία εκατομμυρίων ανθρώπων. Όμως εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο έχει την δυνατότητα, παρουσιάζει εγγενώς το δυναμικό να προκαλέσει ζημία. Αλλά τι να σας πω, ε, ε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα και στη δικιά σας χώρα έχουμε ανάκαμψη των εξαγωγών ε, και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η χώρα σας όντως μπόρεσε να δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας. Ίσως όχι εξαιρετικής ποιότητας θέσεις εργασίας, αλλά παρόλα αυτά από το 7% φτάσατε σε 16 ε, ε, συγγνώμη, το ανάποδο από 16% φτάσατε στο 17% ανεργίας και αυτό είναι πολύ καλό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλία. Ε, μετά από την Jobs Act του ε, Πρωθυπουργού Ρέντζη δημιουργήθηκαν εκατομμύρια θέσει απασχόληση. Επομένω, οι μεταρρυθμίσει βοηθούν και οι μεταρρυθμίσει φέρνουν αποτέλεσμα. Να μην ε, κρυβόμαστε πίσω από του εμπορικού ε, πολέμου ε, για να πούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε μεταρρυθμίσει. Όχι, μεταρρυθμίσει και ξανά μεταρρυθμίσει δεν θα το πω ποτέ αρκετές φορές ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Αλλά βεβαίω καλύτερα θα ήταν να μην έχουμε και του εμπορικού πολέμου. Ε, όσον αφορά τώρα τους, ε, ε, τις αμοιβέ, τους ε, ε, η τεχνολογία μπορεί να αποβεί ε, αποτρεπτική όσον αφορά τους ε, μισθούς. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι απειλούνται και λένε ας πάρω μια δουλειά οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή γιατί διαφορετικά μπορεί να μην βρω ποτέ δουλειά. Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Ξέρετε ότι στην Ισπανία ε, έχει αυξηθεί ας πούμε πολύ ο αριθμός των επιθεωρήσεων και των ε, επιθεωρητών ε, για να δούμε ας πούμε αν οι επιχειρήσεις σέβονται τις αρχές και τα συζήτησα αυτά. Θα τα συζητήσω και με τι αρχέ. Μάλλον όχι. Πήγα ήδη την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή, τα συζήτησα με τι Ισπανικέ Αρχέ. Ο κύριο Φραντσούλικα. Τώρα, Υπάρχει συνένεση στον όσα. Υπάρχει όμως μια δέσμη η οποία προτάθηκε Αργεντινή, Ρουμανία, Περού, Βουλγαρία και μια δυσκολία με την Κροατία γιατί υπάρχουν χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν πρόβλημα με την ένταξη τη, λόγω δαφικών προβλημάτων κλπ. Δεν είναι θέματα που αφορούν τον ΩΣΑ ωστόσο. Ε, και βεβαίως έχει ζητήσει και η Βραζιλία να συμμετάσχει, αλλά προς ώρας δεν υπάρχει συνένεση γιατί υπάρχει ακόμα μία χώρα η οποία δεν θέλει να υποστηρίξει την ένταξη της Βραζιλίας. Ε, για τη Ρουμανία υπάρχει συνένεση. Ωστόσο, εάν δεν συμφωνηθεί η δέσμη των έξι, δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Άρα δεν αφορά προσωπικά τη Ρουμανία. Ε, η Ρουμανία έχει γίνει σήμερα αποδεκτή. Είναι μια χώρα η οποία χαίρει συνενέσεως. Ε, ε, να ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία έτσι ώστε ενδεχομένως να γίνει κάποια στιγμή, δηλαδή μέλος του ΟΣΑ. Παρατηρήσει του κ. Φραντζούλικα εκτός μικροφώνου δεν ακούν οι διερμηνείς. Απαντάει ο κ. Γκουρία. Ναι, συμφωνώ, αλλά κύριε Φραντζούλικα λέτε στο παρελθόν ε, ε, είχαμε μια-δυο χώρες, τώρα έχουμε έξι χώρες οι οποίες θέλουν να γίνουν μέλη του ΩΣΑ. Αυτό με κολακεύει, αυτό με ευχαριστεί. Έχουμε την Αργεντινή, είπαμε το Περού, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία. Και προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση και άλλωστε αυτό αποτελεί πολιτική απόφαση των μελών η οποία χρήζει συνενέσεως και δεν μπορεί να γίνει εάν μία χώρα δεν συμφωνεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία αρνητική ψήφο. Αυτή η αρνητική ψήφος είναι ανασχετική και επομένως δεν μπορεί να προχωρήσει η δέσμη. Αυτό ε, που μπορώ να κάνω είναι ε, παρακαλώ εσείς η μία, η μία αρνητική ψήφο προχωρήστε, αλλάξτε ε, συνεννοηθείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε να λυθεί αυτό το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων με τον ΩΣΑ, με εσάς. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Εκτιμούμε ιδιαίτερο τον ΩΣΑ, αλλά και εσάς προσωπικά, την προσωπική, τους την προσωπική σας δουλειά, τη στήριξη που προσφέρεται για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για την ενίσχυση της ανάπτυξης και για ε, την ε, πολυμέρεια την οποία προτείνεται, για το ότι προτείνεται να ακολουθήσουμε την πολυμερή οδό. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Κουρία.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 So, Συνάδελφοι, ερχόμαστε στο σημείο 9 και 10 απαιτήσει προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων. Μα πιέζει ο χρόνο, γιατί στι 11 θα έχουμε τη δημόσια ακρόαση για τι καταχρηστικές πωλήσει χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αυτό με απογοητεύει κάπως γιατί νομίζω ότι τα θέματα μας τώρα στις 10 ε, είναι πιο σημαντικά και δεν θα έπρεπε να τα συμπτύξουμε μέσα σε ένα μεσάωρο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή που θα μιλήσει στη μητρική του γλώσσα. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκφράζω καταρχάς τις ευχαριστίες μου για τις πολυάριθμες τροπολογίες 337 συνολικά για τον κανονισμό και 205 για την οδηγία έχετε καταθέσει σε πολλά σημεία πιστεύω αποτελούν μια πολύ καλή βάση για βελτίωση περαιτέρω της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιτρέψτε μου να επιστρέψω σε ορισμένα σημεία σε λεπτομέρειες. Κατηγορία 2 και 3. Εγώ στη δική μου έκθεση πρότεινα ένα νέο καθεστώς για τις μικρότερες ε, επιχειρήσεις ώστε να είναι πιο ορατές και να αποφύγουμε και το φαινόμενο του γιογιό, δηλαδή να ανεβοκατεβαίνει μια επιχείρηση στη μία ε, στη μία τάξη, τη μία χρονιά και μετά στην άλλη. Για αυτές που βρίσκονται μεταξύ της κατηγορίας 2 και 3. Ε, Κάποιοι συνάδελφοι υποστηρίζουν ε, με τροπολογίες τους που μπορούν να αποτελέσουν μια καλή βάση. Βεβαίως δεν θα πρέπει α, και συμφωνώ σε αυτό εάν για περιορισμένο χρόνο μια τέτοια επιχείρηση έχει τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας 2 δεν θα πρέπει αυτόματα να μπαίνει σε αυτή την κατηγορία, σε αυτό θα συμφωνήσω και μπορούμε πάνω σε αυτά να έχουμε μια, ε, ένα καλή, καλό τελικό έγγραφο για το κομμάτι αυτό, για την κατηγορία 1 ωστόσο αυτές που βγαίνουν από το καθεστώς όσα. Ε, δεν θα ήθελα υπερβολική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής όταν πρόκειται για ίδιους λογαριασμούς ή όταν πρόκειται για έκδοση ε, χρηματοπιστωτικών ε, μέσων στα 5 δισεκατομμύρια. Ξέρω ότι το επιχείρημα είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά είμαι πάντα πολύ επιφυλακτικός υπάρχει λόγος που έχουμε αυτό τον ειδικό κανονισμό για τις ε, ε, εταιρείε αυτές έκδοσης τίτλων ότι ακριβώς δεν είναι τράπεζες. Δηλαδή δεν μπορούμε να τι μεταχειριστούμε σαν να είναι τράπεζες. Ιδάλω δεν χρειάζεται ειδική ε, ρύθμιση. Εν πάση πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνοηθούμε. Το κύριο αίτημα είναι να υπάρχει χρησιμότητα σε έναν τέτοιο κανονισμό. Μετά έχουμε μία σειρά από τροπολογίες που στόχο έχουν να διευκολύνουν υποτίθεται τις επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα όταν πρόκειται για διευκολύνσεις ή δωρεές, η αποκάλυψη τους δεν νομίζω ότι βοηθά ιδιαιτέρως. Ε, ούτως ή άλλως θα μπορούσε να καλύπτεται αυτό από, τις λιπές από τη λυπή νομοθεσία. Μετά, θέματα τα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερο, όπως το περιβάλλον. Θα μπορούσαμε αυτά να τα συζητήσουμε περισσότερο. Έχει η Επιτροπή στοιχεία ορίσει, ε, τα οποία θα πρέπει να μην αποκαλύπτονται εφόσον δεν έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα για τον ε, καταναλωτή ή επενδυτή. Μπορούμε σε αυτό να συμφωνήσουμε. Εδώ θα έρθω στο θέμα της ε, απόσβεσης όταν είναι μεταβλητή και επιτρέπει την ε, ασφάλιση ωφελών για τον επενδυτή είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Βέβαια στα αξιόγραφα δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαμε σε σχέση με τις τράπεζες σε σχέση με τη δυνατότητα να φορολογείται η διαχείριση των, ε, του ενεργητικού. Εδώ δεν υπάρχει επίδραση στην ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη ε, παρέμβαση καρονιστική στο θέμα της αποζημίωσης σε σχέση με, την, με τις αποφάσεις που έχουν ε, σημασία για την ανάληψη κινδύνου. Επίσης θα πρέπει να δούμε τα κριτήρια ισοδυναμίας, οργάνωση προβλέψεων, και συμπεριφορά στάση, αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το έχουμε στον κανονισμό μας, έτσι ώστε οι ε, εταιρείε αυτές τρίτων κρατών να έχουν αντιμετώπιση ισοδύναμη με αυτήν που έχουν οι ευρωπαϊκές. Ευχαριστώ τους αδέλφους για την υποστήριξη, με τις τροπολογίες τους που όμως μερικές φορές παρά είναι λεπτομερείς και υπησέρχονται σε τομείς της ΜΥΦΙΤ 2. Νομίζω ότι εκεί θα αρκούσε να έχουμε μόνο μία παραπομπή. Και στην ε, ισοδυναμία πρέπει να αφήσουμε ένα περιθώριο, όπως το έχουμε άλλωστε πολλές φορές πει, ε, ε, επιλογών και διακριτικής ευχήρης ε, και της αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, εάν θα πρέπει η OTF και η MTF τρίτων κρατών να απαγορευτούν τελείως, είμαι κάπως επιφυλακτικός, θα έπρεπε να υπάρχει κάποια λογική πρόταση Βεβαίω και μπορούμε να έχουμε μια πιο αυστηρή προσέγγιση σε σχέση με τα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μπορούν οι συνάδελφοι με τα επιχείρηματά τους να με πείσουν. Στις αποφάσεις για την ε, ισοδυναμία, για το αν θα πρέπει να είναι ε, κατά εξουσιοδότηση πράξεις ή εφαρμοστικές. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ε, λόγος να είναι απλώς εφαρμοστικές. Υπάρχει ε, ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί, άλλωστε το έχουμε συζητήσει και με το ευρωπαϊκό, με το αμερικανικό και καναδικό σύστημα Με χαρά βλέπω ότι και οι πράσινοι με υποστηρίζουν. Οι τροπολογίες εν όλο αποτελούν μια γερή βάση για περαιτέρω συζήτηση. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση σκιωδών συγητών στο Στρασβούργο, προβλέψει και πιστεύω ότι μπορούμε τα διάφορα στοιχεία και οι factors κτλ. να τα, key ε, κτλ. να τα δούμε ε, πολύ γρήγορα για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα από τη συνεργασία αυτή. Ευχαριστώ. Ε, τέλειωσε ο εισηγητής και λαμβάνουν το λόγο οι σκιώδεις. Μάντι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω και εγώ να εκφράσω τη στήριξή μου στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ισορροπημένη πρόταση, τεχνικός άρτια και θα πρέπει να διατηρηθεί. Γι' αυτό και δεν στηρίζω τις τροπολογίες συναδέλφων που επανεισάγουν περισσότερα στοιχεία ε, του RR και του CRD σε αυτή τη νομοθεσία. Πράγματα που έχουν σχεδιαστεί για τις τράπεζε και δεν μπορούν να συμπεριλάβουν τους κινδύνους που προκύπτουν από το διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθούν οι επενδυτικέ επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να καλύψουμε τις μη συστημικέ επενδυτικέ επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, δεν στηρίζω τις τροπολογίες των συναδέλφων που προτίθενται να αποδυναμώσουν τα προαπαιτούμενα για την κεφαλαιακή επάρκεια και που θέλουν να αλλάξουν τα κατόφλια για όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στην κατηγορία 3. Θεωρώ την αρχική πρόταση αρκετά ισορροπημένη και βεβαίως ε, επιδέχεται βελτιώσεων. Για τους ε, και factors σωστή αναλογική προσέγγιση για την κάλυψη του παράγοντα κινδύνου, μπορούμε να έχουμε μικρές αλλαγές για καλύτερο υπολογισμό και καλύτερη αποτελεσματικότητα. Και γι' αυτό παρουσιάζουμε τροπολογία να αυξηθεί σε ένα χρόνο η περίοδο για τον υπολογισμό των ημερήσιο του trading. Και τέλος θέλω να αναφέρω και το θέμα της αμοιβή και της διακυβέρνησης, της διαχείρισης, το remuneration και governance. Δεν στηρίζω την ευθυγράμμιση με το καθεστώς CRR και CRT. Οι βασικές αρχές για την αμοιβή και την διαχείριση και τη διοίκηση που ισχύουν για το πιστοτικό τομέα, για το τραπεζικό τομέα, πρέπει να ισχύσουν και εδώ. Τα κίνητρα για τους trader δεν θα πρέπει να είναι ε, μόνο ε, το πρόθεσμο κέρδος, κάτι το οποίο βάζει τους πελάτες τους σε κίνδυνο και γι' αυτό και την διάτα... Ε, τη διάταξη της Κομισιόν και προτείνω την αναδιατύπωσή της. Να επιμείνουμε στο θέμα της ισότητας του φύλου, της ισορροπίας εκπροσώπησης μεταξύ των δύο φύλων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μου. Η αμοιβή τους να είναι ουδέτερη από πλευράς φύλων. Στηρίζω τα μέτρα διαφάνειας της πρότασης αυτής. Reporting αναχώρα το Κοινοβούλιο ανέκαθεν ήταν υπέρ των, της δράσης για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και γιατί ορισμένοι συνάδελφοι να διαγράψουν αυτές τις διατάξεις εδώ. Αυτό με εκπλήσει. Και δεν γίνεται και αναφορά στη, στη βιώσιμη χρηματοπιστωτική, στη, στα θέματα ε, του περιβάλλοντος, στην μια διοίκηση εικον, περιβαλλοντικός φιλική. Να συμπεριλάβουμε αυτά που έχουμε ε, γράψει ήδη στην έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Άρα είναι πολύ τεχνικός αυτός ο φάκελος, παραμένουν κάποια ζητήματα εκκρεμή και πολύ φοβάμαι δεν θα είμαστε σε θέση να τα λύσουμε σε αυτό το στάδιο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όταν αρχίσουν να ισχύει η νομοθεσία αυτή θα φανούν τα προβλήματα. Άρα γι' αυτό και εγώ έχω υποβάλει τροπολογίες για τη ρήτρα αναθεώρησης, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την συμβουλευτική. Οι κανόνες για την εφερεγγιότητα και για το κατακαιρματισμό, για το διαχωρισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων δεν είναι κάτι που είναι πολύ σαφές να ευχαριστήσω τον εισηγητή και ε, με χαρά θα συνεργαστούμε στις ε, συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Εσείς θα μιλήσετε εκ μέρους του Αρμοδίου. Παρακαλώ. Κύριε Στερμπάντη. Ναι, ο κύριος Λούκε δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Ε, στη συγγνώμη και σας διαβάζω τις παρατηρήσεις του. Η πρόταση κανονισμού και οι τροπολογίες του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών δείχνουν ότι υπάρχει ευρύτατη συμφωνία ως προς τη στοχοθέτηση αυτής της νομοθετικής διαδικασίας. Οι επενδυτικές εταιρείες θα πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες μορφές ρυθμίσεις με αυτές στις οποίες υπαγόνται οι μεγάλες τράπεζες όταν είναι συστημικής σημασίας. Μικρές επενδυτικές ε, ε, εταιρείε ή μεγαλύτερες χωρίς όμως συστημική σημασία δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν ε, κινδύνους θα πρέπει να έχουν δραστηριότητα σύμφωνα και με το ποσοστό κινδύνου. Η αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως προς το εύρος και το βάθος της νομοθετικής παρέμβασης. Ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Ε, παραδείγματι θα πρέπει να συζητήσουμε πόσο προσήκον είναι να δίνουμε οδηγίες λειτουργίας σε επενδυτικές τράπεζες που δεν έχουν συστημική σημασία και που σε περίπτωση πτώχευσης δεν θα έχουν μεγαλύτερες συνέπειες για την οικονομία από ότι η πτώχευση μιας άλλης μη χρηματοοικονομικής ή επενδυτικής μεγάλης, ε, ή μεγαλύτερης επιχείρησης. Επίσης συζητούμε εάν η τάξη των μικρότερων και μη δικτυωμένων επιχειρήσεων ε, που ε, περιγράφεται ως υπερβολικά μικρή αντιμετωπίζει φραγμούς τελικά για ε, πρόσβαση στην αγορά που απαγορεύει οδηγούν στην απαγόρευση κάθε δραστηριότητας το νομοθέτημα όπως προτείνεται στηρίζεται πράγματι σε μια αντικειμενική αξιολόγηση και πρόληψη κινδύνου ή τελικά απλώς ενισχύει την ανταγωνιστική ή μάλλον υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα ορισμένων επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους ένταξη στην αγορά. Η παροχή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις αξιογράφων πρέπει να προσφέρεται κατά τρόπο αντικειμενικό και διαφανή Απαραίτητη είναι η πρόνοια για την αντιμετώπιση και πρόληψη του κινδύνου κατά τρόπο αντικειμενικό. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σημασία ή δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση του κινδύνου ή στην πρόληψη αυτού, δεν θα πρέπει να περιορίζονται στη δράση τους. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία με τον εισηγητή και τους εκπροσώπους των λοιπόν ομάδων στις προσεχείς εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος. Ευχαριστώ και ελπίζω να μπορέσει να έρθει. Ναι, βεβαίω βεβαίω ε, στις συνεδριές των σκιωδών. Φιλελεύθερη. Τόρβαλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν την ε, διαβάσουμε, βλέπουμε ότι ενσωμάτωσαν τις συμβουλές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, της EBA. Και άρα αυτό με δύο λόγια μας δείχνει τους τομείς τους οποίους πρέπει να δουλέψουμε, που πρέπει να βελτιώσουμε. Διότι αν δούμε τα πράγματα από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, να πούμε εντάξει, αυτοί ασχολούνται με τη χρηματαγορά και αν δεν είναι τράπεζες, δηλάρουν και κάνουν trading σαν τράπεζες, άρα να ρυθμίζονται ως σαν να τράπεζες σαν να επρόκειτο περί τραπεζών. Όμω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε υιοθετήσει κάπω διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα. Βλέπουμε ότι οι επενδυτικέ επιχειρήσει δεν είναι τράπεζε και δεν θα έπρεπε να ε, υπάρχουν κανόνε που να τι αντιμετωπίζουν σαν να ήταν ακριβώ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες. Και άρα γύρονται κάποια ενδιαφέροντα ερωτήματα από την πλευρά μα. Εάν εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση του συναδέλφου, βλέπουμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι καλό, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι βαβαρός σήμερα. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Είμαι βαβαρός από τότε που ο Ναπολέοντας μας έκανε βαβαρούς. Βαβαρός ή βάρβαρος, τι ακριβώς είπατε. Όχι, δεν είπα βάρβαρος, είπα βαβαρός. Καλώς. Τέλος πάντων, το βασικό ζήτημα είναι αυτό που είπε ο ίδιο ο Μάρκος, δηλαδή πώς χωρίζουμε τις διάφορες ομάδες, τις διάφορες κατηγορίες, ποια κατόφλια θα ισχύουν για την καθεμία. Αυτό το αποτέλεσμα γιογιό που κάνει μια επιχείρηση να πηγαίνει από τη μία κατηγορία στην άλλη. Και άρα επανερχόμαστε στους key factors, οι k factors. Άκουσα τις επικρίσεις. Και κλείνω προς την άποψη του εισηγητή, αλλά όχι, δεν το πάω τόσο μακριά. Για τον κίνδυνο καθαρής θέσεις, για τις εγκυρίσεις, για το clearing. Πρέπει να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς για αυτά τα ζητήματα και τελικά να καταλήξουμε σε μια έκθεση που μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε και στη συνέχεια από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα αυτού του θαυμάσιου οικοδομήματος. Με αδειμονία περιμένω τη συνεδρίαση στο Στρασβούργο να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βεν Κίγκολτ για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, είδατε από τις τροπολογίες μας ότι δεν αποκλίνουμε και τόσο από τη γενική γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του εισηγητή. Ωστόσο, έχουμε κάποια θέματα που θέλουμε να γύρουμε. Δηλαδή, ε, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για το ρόλο και την οικονομική ισχύ που έχουν αποκτήσει ορισμένοι διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού που έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλοι και ξεπερνούν τα στοιχεία ενεργητικού που ε, διαχειρίζονται τα 100 δις, η BlackRock για παράδειγμα και διάφοροι άλλοι τέτοιοι. Αυτοί επηρεάζουν λοιπόν την οικονομία μας, διότι διακρατούν πολύ σημαντικά τμήματα του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού των μεγάλων επιχειρήσεων, όχι μόνο στη γερμανικών, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν απαγορεύεται βέβαια αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες διαφάνειας, έτσι ώστε η κοινή γνώμη να έχει μεγαλύτερο λόγο και να έχει και καλύτερη άποψη για το τι ζητούν αυτοί οι διεθνείς επενδυτές. Τα συνδικάτα, η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας ενδιαφέρονται ιδιαίτερως για αυτό το θέμα και πρέπει να πούμε ότι έχουμε υψηλότερες υποχρεώσεις για τους πολύ μεγάλους παίκτες και πιο αναλογικούς κανόνες για τους μικρότερους παίκτες. Αυτό είναι σαφές. Δεύτερον, συμφωνούμε με τους σοσιαλιστές μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δούμε τις αποκαλύψεις και υποχρεωτικές δημοσιεύσεις πληροφοριών για θέματα, επίσης το θέμα της φορολογίας και της μεταβλητής αμοιβή. Ο λόγος για τους οποίους έχουμε αυτούς τους κανόνες για την αμοιβή των διαχειριστών δεν είναι μόνο αυτός που νομίζετε και το λέω αυτό σε σύνδεση και με τους ε, εκπροσώπους από το ECR και τα λοιπά. Είναι πρόβλημα και για, τα συστημ, για τις συστημικό σημαντικές επενδυτικές επιχειρήσεις. Καλλιεργείται ένα κλίμα και μια κουλτούρα σε αυτό το κλάδο της οικονομίας που τελικά απειλεί ε, την οικονομία Δηλαδή είναι κανόνες ανταμοιβή που βασίζονται στο short-term selling, στις βραχυπρόθεσμες πωλήσει, στην σημείωση κερδών σε βραχυπρόθεσμη βάση, ε, προκυκλική αντιμετώπιση από πλευράς οικονομικής θεωρίας, κάτι το οποίο ε, τους κινεί να, ε, να αγοράζουν περισσότερο και να πολλούν τέτοια προϊόντα και γι' αυτό έχουν υψηλότερη ανταμοιβή καλλιεργείται ένα κλίμα και μια κουλτούρα δηλαδή η οποία είναι δυσάρεστη και θέλουμε εμείς να αλλάξει αυτή η κουλτούρα προς μια πιο βιώσιμη αντιμετώπιση σε βάθος χρόνου, μακροπρόθεσμα δηλαδή. Η... Οι φορολογικοί κανόνες δεν είναι η σωστή βάση για να επιβάλλουμε την αρχή της αναλογικότητας. Έχουμε μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση, αυτό θέλουμε. Και άρα οι επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να κάνουν reporting αναχώρα δεν είναι οι μεγάλοι παίκτες. Γιατί συνήθως υπάρχει μία έδρα όπου ασκείται μία επιχειρηματική δραστηριότητα στους μικρούς παίκτες Άρα το reporting αναχώρα είναι ένας τρόπος να είναι πιο δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν έδρα σε μία χώρα και μία μόνη έδρα και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε πολλά και διαφορετικά κράτη. Δεν είναι αυτά παιδεία για να εφαρμόσουμε την αναλογικότητα, αλλά να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Συμφωνούμε και με τη διάσταση του φύλου. Δεν υποβάλαμε τροπολογίες για τον παράγοντα K. αλλά θέλουμε να αποφύγουμε τη διαιτησία. Και συμφωνούμε με αυτές τις τροπολογίες. Συμφωνούμε και με τις τροπολογίες του κ. Βέρνερ Λάγκε. Να έχει μεγαλύτερη επιρροή η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και όχι τόσο μεγάλη η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Και θα πρέπει να επανεξετάσουμε το κατόφλι των 30 δις και να το ορίσουμε καλύτερα. Αυτά λοιπόν από την πλευρά μας και θα λειτουργήσουμε επικοδομητικά, να βρούμε συμβιβασμούς, περιμένουμε τις συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ, Μιγγέλ, για την ΚΟΕ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η πρόταση στην ουσία επανέρχεται σε αυτή την ε, αγορά, την ε, ε, κεφαλαιακή αγορά που δίνει δυνατότητα χρηματοδότησης ε, των επιχειρήσεων μέσω προσέγγισης ευρωπαϊκών κανόνων με τόσο συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Και επανέρχομαι σε μια ερώτηση η οποία υπευλήθηκε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑΜΑ. Γιατί οι επενδυτές δεν, δεν επιλέγουν αυτήν την οδόμα, γιατί υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές ανάμεσα στους επενδυτές των χωρών και εμείς δεν υποστηρίζουμε με αυτήν την ε, ιδέα ε, ε, υποχρέωσης θέσπισης κανόνων και κανονισμών που, θα, που θα υποβηθούν τις εταιρείε. Μα εάν δεν ενεργήσουμε με τον τρόπο αυτό, τότε οι επενδυτές ίσως θα μπορούσαν να απαντήσουν οι ίδιοι στα ερωτήματα αυτά. Εγώ πάντως αναρωτιέμαι εάν πραγματικά θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των επιχειρήσεων Λοιπόν, γιατί οι όροι που αναφέρονται εδώ με προβληματίζουν. Υπάρχουν και κά... Υπάρχει και κάποια άλλη ερώτηση που δυστυχώς δεν μπορώ να μην ε, αναφέρω. Εάν ε, υφίσταται συστημικός ε, κίνδυνος, εδώ μιλάμε για τα λεφτά των φορολογούμενων πολιτών. Εάν λοιπόν υπάρχει συστημικός κίνδυνος, αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε το ε, ενδεχόμενο δυνατότητας αντιμετώπισης αυτού του συστημικού κινδύνου με εναλλακτική την χρήση δημοσίου χρήματος προς αποφυγή καταστροφής που εάν επέρχεται θα ήταν ε, πολύ ε, μεγαλύτερος. Τώρα, εάν δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος δεν χρειαζόμαστε τέτοια διευθέτηση, τέτοιο κανονισμό το θέμα της της, ε, του υπερβολικού κινδύνου ε, ναι, μας ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι η κάλυψη του φορολογικού κινδύνου είναι κάτι απαραίτητο και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και στις, στις εκθέσεις αναχώρα και το θέμα της ισότητας των φίλων επίσης είναι πολύ καλό. Λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχει άλλος συνάδελφος που να θέλει το λόγο από το ΙΕΝΕΦ e ή από το EDTF. Ωραία, είμαστε στο Catch the Eye επομένως. Merci. Η Άννα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε. Εγώ Δυστυχώς ε, ήμουν σε άλλη συζήτηση, λέει η κυρία Σαντέρα, και δεν ε, μπόρεσα να είμαι εδώ από την αρχή. Ωστόσο, ε, πρώτα θα ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του, αλλά θέλω να υποβάλω δύο ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, ο διαχωρισμός ανάμεσα στην τάξη 1 και την τάξη 2. Η τάξη 1 που προτείνεται από την Κομισιόν φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένη Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες ε, έχουν bank-like δραστηριότητες ε, και που μπαίνουν στο, στην τάξη 2 λόγω ε, του προϋπολογισμού, του ισολογισμού συγγνώμη, 30 δις που κρίνεται πολύ υψηλός και επομένως θα μπορούσαν να είχαν και επομένως μπορούν να έχουν περιορισμένο εποπτικό έλεγχο ενώ παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο. Πιστεύω ότι αυτή η έννοια του κατοφλίου θα πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει να πέσει το κατόφλι. Δεύτερον, ο καθορισμός των ισοτιμιών. Εδώ υπάρχει το σύστημα της φυσικής ε, παρουσίας μέσω θυγατρικής ε, ή... Ε, concurrence ε, ή υποκαταστήματος ε, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διαφετηθεί γιατί υπάρχουν ε, επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να υποχρεωθούν να φέρονται ως ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και επομένως δεν θα πρέπει απλώς να αφήσουμε στα χέρια των αρχών της τρίτης χώρας τη διαδικασία ελέγχου της ευρωπαϊκής συμπεριφοράς και επομένως ε, η άμεση απευθείας επιθεώρηση, επιτήρηση από την ΕΣΜΑ πιστεύουμε ε, και αυτών των θηγατρικών ε, κλπ παραμένει ο καλύτερος τρόπος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, δεν έχω άλλον στον κατάλογό μου για το Κάτσο αδειά ή θέλει μήπως Θέλει μήπως η Κομισιόν να πει κάτι, όχι από ό,τι φαίνεται δεν επιθυμεί. Ε, επομένως ε, εσείς επαφίεστε στη σοφία μας. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια και θα δώσω το λόγο ε, στον εισηγητή, ο οποίος θα ξαναπάρει το λόγο στη μητρική του γλώσσα. Και σας ευχαριστώ θερμά για τις παρεμβάσεις σας μπορούμε να έχουμε νομίζω μέσα στο φιλοδόξο, φιλόδοξο χρονοδιαγράμμα που έχουμε ορίσει και που πρέπει να είμαστε θέση να τηρήσουμε ένα καλό κείμενο έτσι ώστε αυτό το νομοθετικό πακέτο με τον κανονισμό και την οδηγία να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητεία ε, με τις διαπραγματεύσει του Συμβούλου και την έγκριση βέβαια. Αυτός πρέπει να είναι ο κοινός μας στόχος. Δεν ναι, θα επισέλθω στις διάφορες ε, λεπτομέρειε Στην επιμέρειες σημεία απλώς. Ένα ζήτημα το οποίο με κατέπληξε και ήθελα να το επισημάνω, με ξαφνιάζεται ότι μια κυβέρνηση που δεν έχει κανένα βουλευτή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταφέρει να βρει τόσους πολλούς υποστηρικτές μέσα στην Επιτροπή μας που διατυπώνουν τις σχετικές τροπολογίες. Θα το κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή λοιπόν. Η Εποπτική Αρχή της εν λόγω χώρας με έχει συναντήσει, έχουμε συζητήσει, έχουμε ασχοληθεί με πολλά σοβαρά ζητήματα και έχουμε πάνω απ' όλα σταθεί στο τι είναι τράπεζα, τι είναι επενδυτική επιχείρηση, ποια είναι η διαφορά ανάμεσά τους. CRD, CIR και τι μπορεί να ισχύσει και για τις επενδυτικές επιχειρήσεις μια σειρά από επιχειρήσεις που ρητά μάλιστα αναφέρθηκαν εδώ θα έπεφταν στην κατηγορία 1 και άρα θα πήγαιναν στο CRD, CIR. Και άρα νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πώς θα τα διαμορφώσουμε αυτά και πώς θα ορίσουμε τα όρια και τα κατόφλια για την υπαγωγή στην τάξη αυτή. Οπωσδήποτε είναι ενδιαφέρον να δούμε και το ότι υπάρχει τόση πολλή κινητοποίηση και το τι αποτέλεσμα μπορούμε να φέρουμε. Κάτι άλλο βέβαια που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ο κίνδυνος. Ποιος αναλαμβάνει το κίνδυνο στις ε, συστημικά σημαντικές ε, τράπεζες και τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ενισχύθηκε αυτό. Ορίστηκε μια ιεράρχηση δομών πιστωτών με απαλλαγή από την υποχρέωση για τον φορολογούμενο να συμβάλλει οικονομικά, για τις επιχειρήσεις, τις επενδυτικές δεν ήξερα, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν υπήρχε. Όχι, μα νομίζω. Έχω το δικαίωμα να ομιλώ, λέει ο πρόεδρος και η συγητής Ακούστηκε κάποια φωνή από την αίθουσα. Υπάρχει λοιπόν εν τέλει κίνδυνος τον οποίο αναλαμβάνει ο φορολογούμενος για τις επενδυτικές αυτές επιχειρήσεις ή όχι όλα αυτά που είναι και επώδυνα και λυπηρά. Δεν πρέπει να καλύπτεται βέβαια ο κίνδυνος αυτός, όσο δύσκολο και αν είναι, από τον τελικό πιστωτή, το φορολογούμενο. Ως τελικό πιστωτή από το φορολογούμενο. Ίσως θα πρέπει όταν έχουμε μια διαχείριση ενεργητικού ο, και ο διαχειριστής αναλαμβάνει μια στρατηγική ε, για τους επενδυτές του, από την οποία θα ωφεληθούν. Δεν θα πρέπει και αυτό σε περίπτωση ε, που κάνει κάποιες ασφαλμένες επιλογές να ενέχεται σε ένα βαθμό έστω. Επομένως, ε, διαφάνεια μπορούμε να έχουμε και από την αγορά ούτως ή άλλως και πέραν της ρυθμιστικής μας παρέμβασης. Ε, θα, είναι ότι η συζήτηση που θα έχουμε από κοινού θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και βέβαια είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και επικοδομητικό κλίμα συνεργασίας με τους και οδησηγητές των ομάδων. Μπορούμε να αρχίσουμε αυτή τη δουλειά για να έχουμε ένα συμβαστικό κείμενο έτοιμο εγκαίρος πάνω στο οποίο θα εξασφαλίσουμε ελπίζω συμφωνία. Εγώ πάντως θα κάνω ό,τι μπορώ ε, στο βαθμό της, ε, των δυνατοτήτων μου είτε για να συνεργαστούμε στο δυνατόν καλύτερα. Τώρα προχωράει ο χρόνος και μια και τέλειωσε την παρουσίασή μου ως ηγητής. Ε, γυρνάω στα αγγλικά και πάλι, έχουμε κερδίσει λίγο χρόνο <clears throat> για το επόμενό μας θέμα. Είμαστε τέσσερα λεπτά μπροστά. Α, ναι, όχι, ξαναγυρνάω στην έκθεσή μου και το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, προθεσμία για τροπολογίες είχε κλείσει, αλλά την παρατείναμε κατόπιν αιτήματος μίας ε, ομάδα στην Οικονομική Επιτροπή προβλέπεται προς το παρόν να ψηφιστεί στις 24 Σεπτεμβρίου εάν προλάβουμε βεβαίως και με την διαπραγματευτική ομάδα να κλείσουμε το θέμα ή τέλος θα δώσουμε ένα, μικρότερο περιθώριο, ένα μικρό ακόμη περιθώριο. Πάντως θέλουμε πριν από το τέλος του χρόνου να γίνει η θελω να δωσουμε ενα μικροτερο περιθωριο ενα μικρο ακομη περιθωριο παντως θελουμε πριν απο το τελος του χρονου να γινει η ψηφοφορια στην Επιτροπή στο, στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί παράλληλα με τη διαδικασία του Συμβουλίου και να πάμε στους τρεμερούς διαλόγους αν όχι υπό Αυστριακή, πάντως υπό Ρουμανική Προεδρία. Καλώς, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό ε, διάλειμμα. Ενημερώνομαι ότι θα έρθει πάλι ο Πρόεδρος μας, ο κ. Γκουαλτιέρη, αλλά όπως και να έχει, στις 11 θα ξεκινήσουμε. Respond. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από το μικρό αυτό διάλειμμα, ο πρόεδρος μας κάνει διαπραγμάτευση με έναν από τους ε, ομιλητές. Θα πρέπει ωστόσο να κάνουμε να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά μας για την καταχρηστική πώληση των ε, οικονομικών προγραμμάτων. Η ε, συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο και παρακαλώ να ξέρετε ότι όλος ο κόσμος μας παρακολουθεί. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε μια σειρά από προϊόντα που έχουν εμφανιστεί πρόσφατα τα τελευταία χρόνια Εν τω μεταξύ, οι διερμηνεί σα ενημερώνουν ότι η εργασιακή διαμάχη που οφείλεται στη μονομερή επιβολή συνθηκών εργασία μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα. Έχουν ε, επιστρατευτεί συνάδελφοί μα από ε, ορισμένε καμπίνε και σε ένδειξη διαμαρτυρία ε, και αλληλεγγύη προ αυτού, εμεί συνεχίζουμε να δουλεύουμε και δεν προβαίνουμε στη στάση εργασία που είχε ανακοινωθεί, καθώ δεν θα ήταν ισότιμη μεταχείριση για όλου του διερμηνεί. Και συνεχίζουμε. Θέλουμε λοιπόν να κοιτάξουμε τα θέματα της καταχρηστικής πώληση, ε, να αντιληφθούμε το ρόλο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην υπόθεση αυτή, MIFIR, MIFID, IFD, USITS. Καταρχάς, καλό τους ομιλητές μας στο βήμα. Έχετε από πέντε λεπτά. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. ερωτήσεις και αποκρίσεις με δύο λεπτά για τους, ομιλητές, για τους ε, ερωτώντες βουλευτές και τρία για τους ε, ομιλητές μας. Ο κύριος Φλάβιο Μποντζοβάνη από την Κόνσοπ της Ιταλίας, η κυρία Μπεναχάινα από την Beta ο κύριος Σέξπι από από το Τμήμα Προστασίας Καταναλωτών ε, της ε, ΑΙΟΠΑ, ο Τίλμαν Λούιτα, γνωστός και μη εξαιρετέως εδώ, της μονάδας τραπεζικών αξιών και τίτλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε ακόμα και τον κύριο που εκπροσωπεί την ΑΕΜΕΦ τη Γαλλία ο Τωρίτιο ε, ο οποίος έχει κατηδίαν συστήσει με τον κύριο Γουαλτιέρη αυτή τη στιγμή. Ε, ξεκινώ λοιπόν αλλάζοντα τη σειρά και καλώντα τον κύριο Φλάβιο Μποντζοβάνι ε, να ξεκινήσει πρώτο. Σα ευχαριστώ που, καλε, που δεχθήκατε την πρόσκληση. Έχετε το λόγο κύριε Μποντζοβάνι Χωρί μικρόφωνο κύριο Μποντζοβάνι δεν ακούνε οι Παρακαλώ πιέστε το, ανοίξτε το μικρόφωνο σας γιατί δεν σας ακούμε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που δίνετε στην Κονσόμπ, την οποία εκπροσωπώ, ε, να δώσει την συμβουλή της όσον αφορά ε, το mis-selling των ε, προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό των διαθεσίμων πόρων, είναι απαραίτητη η κάθε αρχή προληπτικής εποπτείας με τρόπο διαρθρωμένο και αντικειμενικό να ασκεί τις δραστηριότητες επιτήρησης. Ε, οι προτεραιότητες και η επιλογή της τυπολογίας τους ε, θα πρέπει να ακολουθεί μία λογική βασισμένη στον ε, κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες, διαθέσιμους πόρους κλπ. Το μοντέλο επιτήρησης το οποίο προτείνει η Κόνσομπ λαμβάνει υπόψη την περιοδική αναέτηση έτος ε, έκθεση όσον αφορά ε, τις ε, τράπεζες. Επίσης, διαρκή επιτήρηση όσον αφορά τις τράπεζες οι οποίες έχουν πάνω από 80% της εγχώριας αγοράς, καθώς επίσης και ένα σύστημα ποσοτικής αξιολόγησης βάσει του σχετικού κινδύνου που παρουσιάζουν οι τράπεζες όσον αφορά τη μη συμμόρφωση. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν αυτό το μοντέλο προκύπτουν και διάφορες ε, άλλες ε, διαδικασίες επιθεώρησης ε, που αφορούν ακριβώς το enforcement καθώς επίσης και τις κυρώσεις. Λαμβάνονται υπόψη επίσης και οι αρχές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της ΕΣΜΑ. Όσον αφορά την CONSOB, η οποία, είναι, η οποία ασχολείται με και είναι υπεύθυνη για την προστασία των επενδυτών και τις δράσεις των τραπεζών ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε το Mrs. Selling να μας ε, απασχολήσει ιδιαίτερα αυτές δηλαδή οι καταχρηστικές ε, πωλήσει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη και οι, οι πελάτες λιανικής. Μετά από την δημιουργία της BRRD συγκεκριμένες έρευνες έχουν γίνει και αναλύσεις όσον αφορά κυρίως τον εσωτερικό έλεγχο των μεσαζόντων ε, κυρίως ε, ε, με το μοντέλο υπηρεσίας Tide Agent. Υπάρχουν επίσης γίνει πάρα πολλές δράσεις επιτήρησης και έχουν επιβληθεί πολλές, πολλά διοικητικά πρόστιμα κυρίως για δραστηριότητες μεταξύ του 2011 και του 2015. Επίσης έχουν προχωρήσει αρμοδίως προς ε, τις ποινικέ διαδικασίες ορισμένες ε, ε, ειδικέ περιπτώσεις. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν πολλές φορές συγκρούσεις συμφερόντων οι οποίες δεν διαχειρίζονται σωστά και δεν δηλώνονται σωστά. Θεωρούμε επίσης ότι υπάρχουν δραστηριότητες και δράσεις οι οποίες, οι οποίες εκφεύγουν τις MIFID. Το 2017 Ευχαριστώ. Οι ε, ενδιάμεση που έχουν ε, ε, υποστεί κυρώσεις από την Κόνσομπ ήταν στον αριθμό 15. Επίσης έχουν υπάρξει εμπλοκές με 282 επιχειρήσεις και τα πρόστιμα έφτασαν στα 11,8 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα με τις δραστηριότητες ενδυνάμωσης και επιβολής η Κόνσομπ έχει, έχει δημοσιεύσει και κάποιες ανακοινώσεις ε, οι οποίε αναφέρονται κυρίως σε αυτόν τον κίνδυνο των καταχρηστικών ε, πωλήσεων, ε, της προώθησης προϊόντων αήλων, καθώς επίσης και περιπλόκων μεταξύ των οποίων και ομόλογα subprime, καθώς επίσης και για τους ε, για τους ε, ε, πελάτες λιανικής. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα bail-enable προϊόντα. Επίσης έχουν καταδειχθεί οι βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Ε, μέσω αυτών των διαδικασιών και μέσω του soft law ε, το Ινστιτούτο έχει προχωρήσει σε σημαντική μείωση ε, των εγχωρίων χρηματοπιστωτικών προϊόντων υψηλού κινδύνου για τους πελάτες λιανικής. Πρέπει να πούμε ότι οι περιπτώσεις self-placement έχουν μειωθεί από 320,4 δις ευρώ, δηλαδή 1,4 του συνολικού ε, το Δεκέμβριο του 2011 στο 95,6 δις ευρώ, δηλαδή 9,94 του συνόλου των χρηματοπιστωτικών προϊόντων ισχύρας ε, πελατών λιανικής το Σεπτέμβριο του 2017. Επίσης, από την 9η Ιανουαρίου του 2017 έχει θεσπιστεί ε, στην Κόνσομπ ο διαιτητής όσον αφορά ε, τις χρηματοπιστωτικές ε, διαφορές. Στους πρώτους 17 μήνες δραστηριότητας ο διαιτητής έχει μελετήσει 2.542 προσφυγές πρόσφυγε, 700 τους πρώτους 5 ε, μήνες το 2018 μόνο και επίσης έχουν ε, ληφθεί 625 αποφάσεις, δηλαδή 60% μάλιστα ε, των φορών υπέρ του αποταμιευτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάρκο Φέμπερ ήδη έχει καλωσορίσει, λέει ο πρόεδρο Γκουελτιέρη, ε, όλου του ε, Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Ρομπέρτο Φέλπ από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η καταπολέμηση των καταχρηστικών πωλήσεων χρηματοπιστωτικών ε, προϊόντων είναι βέβαια κύριος στόχος μας, ε, όπως και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Χρησιμοποιούμε την ε, εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία ως εργαλεία, αλλά βέβαια κινούμαστε ταυτόχρονα με μια κινητοποίηση σαφέστατη για την, προστασία, για την δημόσια ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και του καταθέτη, αλλά και για την διαπαιδαγώγηση του επαγγελματία. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα από την εμπειρία μας στη Γαλλία το κανονιστικό πλαίσιο έχει ιδιαίτερα εμπλουτιστεί και μας επιτρέπει να καταπολεμούμε καλύτερα τις καταχρηστικές πωλήσει. Παραμένουν ωστόσο ακόμα κάποια κενά που πρέπει να καλυφθούν και αντίστροφα θα επισημάνω ότι πρέπει να προσέχουμε να μην ε, κάνουμε υπερβολική νομοθετική παρέμβαση, γιατί αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό. Πρώτο μήνυμα. Δεύτερο μήνυμα, ε, η παιδαγωγική προσπάθεια είναι συμπλήρωμα απαραίτητο για κάθε κανονιστική και ρυθμιστική παρέμβαση. Πρώτον, λοιπόν, ένα πράγματι ε, αισθητά ενισχυμένο κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Παραμένουν κενά, αλλά πρέπει να προσέχουμε και να μην υπερβάλλουμε στην κανονιστική παρέμβαση. Και εδώ θα πω ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΜΥΦ 2 και ΠΡΙΠΣ έχει, έχει ενισχύσει σημαντικά το πλαίσιο που εφαρμόζεται στην ε, διάθεση στο, ε, στη διάθεση των προϊόντων αυτών που είναι και βέβαια γνωστά και στον και με τα στοιχεία που γίνονται γνωστά στον καταναλωτή. Ιδιαίτερα είναι ενισχυμένοι οι κανόνες σε σχέση με την ε, κοινοποίηση στον πελάτη ε, των στοιχείων ε, του κινδύνου των προϊόντων που πολύ όπω την προβλέπει το MIFID 2. Επίσης υπάρχει ενίσχυση των υποχρεώσεων σε περίπτωση στον τομέα της γνώσης και την ανακύκλωση των προϊόντων, τεκμηρίωση κατάλληλη, υποχρέωση περιγραφής των πακέτων προϊόντων όταν υπάρχει αυτή η περίπτωση, διαφάνεια για τα τέλη ή άλλη επιβάρυνση, για σύγκρουση συμφερόντων. Όλα αυτά ρυθμίζονται. Αλλά πρέπει να προσέχουμε να μην είμαστε και υπερ, ε, υπερβολικά παρεμβατικοί και άρα αντιπαραγωγικοί. Επί παραδείγματι, στα ερωτηματολόγια γνώσεων των... Ε, πελατών πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι υπερβολικά, ότι είναι, παρεμβαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας ή ρωτούν ενοχλητικές ερωτήσεις, Φερρυπίν, αν έχει ενεργητικό που διακρατούν άλλοι διαμεσολαβητές. Πολλές φορές δεν έχουν και μεγάλη σχέση και τελικά παρεμποδίζουν ή αποθαρρύνουν κάποιους από τους εκδότες ή δίνουν πληροφορίες ακατάλληλες μη προσήκουσε. Ιδιαίτερα για τα κοντά, για τα σύντομα προϊόντα. Ή όταν δίνει πληροφορίες για πολύ πρόσφατες επιδόσεις που δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν μελλοντικέ επιδόσεις. Επομένως, μια διαφορετική προσέγγιση θα προτείναμε σε σχέση με τον εκδότη, αλλά και ενθάρρυνση μέσω της νομοθεσίας για διατήρηση ως το δυνατόν μικρότερο αριθμού προϊόντων, να ξεφορτωθεί δηλαδή ο εκδότης τα πιο δύσκολα προϊόντα για να μειώσει και τον κίνδυνό του. Ε, ίσως θα έπρεπε τα επίπεδα 1-2 να περιοριστούν ή και να εκμηδενιστούν και να μείνουμε σε ένα επίπεδο 3 ε, ομοιογενοποιημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κύρια ιδέα ότι επιτρέπουμε την ε, μεγαλύτερη διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκια, δηλαδή προσέγγιση χαρτοφυλακίου πέραν του εις προσέγγισης προϊόντος. Επίσης υπάρχουν ε, ζώνες κινδύνου διάθεσης ε, μη προσήκουσας που δεν καλύπτονται από τους φυστάμινους κανόνες. Φερρυπίν ε, εξουσίες της ε, ΕΣΜΑ σε σχέση με τη δυνατότητα για απαγόρευση ε, προϊόντων, διάθεση προϊόντων που ενέχουν μεγάλο κίνδυνο. Μεγάλη παρέμβαση, έντονη παρέμβαση, την έχει κινητοποιήσει τώρα η ΕΣΜΑ σε σχέση με ορισμένα προϊόντα, Δικά κυρίω αλλά ταυτόχρονα ο προσωρινός χαρακτήρας της παρέμβασης της ΕΣΜΑ ενέχει και τον σπόρο του κινδύου νου ασυνέπεις μεταξύ κρατών για προϊόντα που διατίθενται κατά τρόπο καθαρά διασυνοριακό μέσα πλατφόρμας και δεν δίνει ορισμό για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Ενώ ε, μπορεί να υπάρχουν παρόμοια προϊόντα με χαρακτηριστικά χρηματοπιστωτικών, με αντίστοιχους στόχους, αλλά που δεν καλύπτονται Επί παραδείγματι αυτό που ονομάζεται επένδυση ε, αδάμαντα ή σε κρυπτοενεργητικό. Η εύθυρη παροχή υπηρεσιών δεν ασκείται με αρκετή συμμετοχή των κρατών υποδοχής. Η θέση της πλατφόρμας σε ένα Ευρωπαϊκής Ένωσης με ταυτόχρονη διάθεση σχεδόν όλων των προϊόντων σε άλλα κράτη-μέλη δεν καλύπτεται επαρκώς και οι αρχές του εν λόγω κράτους, του κράτους προελεύσεως δηλαδή, δεν έχουν αρκετά κίνητρα για να παρεύουν στο κράτος ε, της διάθεσης. Άρα δεν υπάρχει αρκετή προστασία. Η διάθεση από τις τράπεζες στους ε, πελάτες λιανικής προϊόντων ε, που διακρατούν με βάση το TILA και το MRAL πρέπει να καλυφθούν από ειδικέ διατάξεις. Και ελπίζουμε ότι με την αναθεώρηση του ε, BRD e θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο μήνυμα. Χρειάζεται η διαπαιδαγώγηση συμπληρωματικά προς την κανονιστική ρύθμιση τόσο για τον επαγγελματία όσο και για τον ιδιώτη. Προσπάθεια που βεβαίως θα αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο αλλά πρέπει να είναι οργανωμένη και στονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως χρειάζεται και να υπάρχει παρακολούθηση και ο έλεγχος της διάθεσης για την ε, προβολή των βέλτιστων πρακτικών και την εκρίζωση των κακών και άρα χρειάζεται έλεγχος εκ των υστέρων έως και εκ των προτέρων και των, ε, των, της πλατφόρμας προστήριξης για τη διάθεση και ανακοίνωση προτεραιοτήτων ε, εποπτείας και θεματική έλεγχη σε σχέση με το αν είναι ο χαρακτήρας των συμβουλών και αν γενικά λαμβάνονται υπόψη και γίνονται σεβαστές οι απαιτήσει της ΜΥΦ 2. Χρειάζεται επίσης να υπάρχουν κύματα ε, ευνίδιων επισκέψεων, ε, μαθήματα που θα πρέπει να διαδίδονται προς όφελος του κοινού, βέλτιστες πρακτικές και μαύρες λίστες δημοσιοποίησή τους πάνω από όλα μέσα από το διαδίκτυο. Επίσης χρήση των μέσων επικοινωνίας, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του facebook, του google, κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να καταγγέλλεται κάθε μη προσήκουσα ε, πρόσκληση ε, προς επενδυτές. Πρέπει επίσης να υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις μέσω πρόθεσμα, παραδείγματι απευθυνόμενες στους νέους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας με την, και την την Τράπεζα ή σε σχέση με το Υπουργείο Εργασίας για τους εργαζομένους ε, που ενδεχομένως θα ήθελαν ε, ή έχουν εμπλακεί σε επενδυτικά σχήματα σε σχέση με την ε, αμοιβή τους. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. να δώσω το λόγο στη Γέλα Μπένερ, πρόεδρο της οργάνωσης Better Finance. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα μιλήσω στα αγγλικά, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε να σας μιλήσω για τις καταχρηστικές πωλήσει χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για όλους τους χρήστες αυτών των προϊόντων που εκπροσωπώ σήμερα ως πρόεδρος της οργάνωσης Better Finance, καλύτερη χρηματοπιστωτική. Κάναμε μια έρευνα πριν από ένα χρόνο για τις καταχρηστικές πωλήσει. Την έχω φέρει την έκθεση και τα πορίσματά της έρευνας. Να τη διαβάσετε αν θέλετε. Είναι ένα ζήτημα που παραμένει και είναι πολύ διαδεδομένο. Οι καταχρηστικές πωλήσει χρηματοπιστωτικών προϊόντων και θα σας δώσω δύο παραδείγματα όπου οι ρυθμιστικές αρχές και οι εποπτικές αρχές δεν έχουν προστατεύσει επαρκώς τους επενδυτές. Ας ξεκινήσω με το PRIPS και το KID, τα Key Information Document, τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για το πακέτο και τον κανονισμό για τα επενδυτικά προϊόντα λιανικής που βασίζονται στις επενδύσεις. Όλα αυτά μπερδεύουν τους επενδυτές. Έχουμε ασκήσει κριτική για τη διατύπωση. Έχουμε μιλήσει για τις αρνητικές συνέπειες που, που έχει εξάλληψη της αναφοράς σε αρνητικές επιδόσεις του παρελθόντος. Τώρα, προβλέψεις μελλοντικών αποδόσεων αυτές που χρησιμοποιεί ο τρέιντερ για να ενημερώσει τους επενδυτές και ο επενδυτής δεν θα ξέρει αν το προϊόν αυτό το χρηματοπιστωτικό έχει φέρει χρήματα στο παρελθόν, πώς θα έχει πάει στο παρελθόν και αν έχει εκπληρώσει τους επενδυτικούς στόχους ή όχι. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία και έχει εξελιχθεί. Ζητούμε ο κανονισμός αυτός για το ΠΡΙΠ να συμπλέει με τους κανόνες της ΜΥΦΙΤ 2 για τις αποκαλύψεις για τις επιδόσεις, ότι δηλαδή οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις μελλοντικέ επιδόσεις θα πρέπει να συνοδεύεται από προειδοποίηση που θα δηλώνει ότι τέτοιου προβλέψεις δεν είναι αξιόπιστος δείκτης μελλοντικών επιδόσεων. Χρειάζεται αναθεώρηση του κανονισμού ε, του ΠΡΙΠ και γι' αυτό θέλουμε να επανεισαχθούν οι πληροφορίες για τη σχετική απόδοση του προϊόντος στο παρελθόν. Η νέα προσέγγιση δεν επιτρέπει στους επενδυτές να συγκρίνουν το κόστος που έχει ένα προϊόν σε σχέση με τα άλλα, με το κόστος των άλλων προϊόντων. Και δεν καταλαβαίνει τον αντίκτυπο των τελών εισόδου και εξόδου. Έχουμε αρνητικό κόστος συναλλαγής και αυτό αποκαλύπτεται στο βασικό πληροφοριακό έγγραφο, στο ΚΙΝΤΕ και άρα δημιουργεί σύγχυση. Θεωρούμε ότι ο αρχικός στόχος του KID, του Key Information Document, είναι να υπάρχει παιχνίδι επίσης όρης και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ζητούμε λοιπόν να υπάρχει αναθεώρηση έγκαιρα στοχευμένη του κανονισμού ΠΡΙΠΕ για αυτή τη χρονιά και επέκταση τριών ετών της εξαίρεσης των κεφαλαίων βάσει του usage. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο παράδειγμα, στο ε, βασικό πληροφοριακό έγγραφο το KID για το usage. Έχουμε έρευνες τις οποίες δημοσιεύσαμε, επικαιροποιημένες, ενημερωμένες, το 30% των ε, βασικών equity fund τύπου usage που έχουν ένα όριο αναφοράς δεν συμμορφούνται με, τις, ε, με τα προαπαιτούμενα για ε, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται, έτσι όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο δηλαδή που αυτά τα ε, ταμεία είχαν νομική υποχρέωση να αποκαλύψουν στοιχεία για το σημείο αναφοράς, για το benchmark που χρησιμοποιηθούν, δεν το έπραξαν αυτό. Και άρα οι ιδιώτες επενδυτές βασίστηκαν σε αυτά τα KID, σε αυτά τα βασικά πληροφοριακά έγγραφα για να λάβουν την επενδυτική τους απόφαση και παραπληροφορήθηκαν ή παραπλανήθηκαν από το μεγάλο μεγάλο αριθμό των KID, των βασικών πληροφοριακών εγγράφων. Η κατάσταση είναι πολύ ανασυχητική. Η οργάνωσή μα έχει δείξει ότι όλα αυτά είναι σε βάρο των ιδιωτών επενδυτών ήδη από το 2017 και έχουμε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών από τότε. Αυτά τα φάντα ε, κυρίως βρίσκονται στο Λουξεμβούργο και στην Ιρλανδία, κατά κύριο λόγο. Αυτά που δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία. Άρα πρέπει να υπάρξουν θέματα και ερωτήματα που να εγερθούν για την επιβολή του νόμου και τις εποπτικές αρχές. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι είναι ανάγκη να βελτιώσουμε τους κανόνες εποπτείας και επιβολής του νόμου και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό. Πρέπει να βελτιώσουμε τη δημόσια εφαρμογή του νόμου, δηλαδή το πεδίο εφαρμογή στη διοίκηση, τη διαχείριση και την αποτελεσματική εποπτεία της ΕΣΑ. Η Better Finance, η οργάνωσή μας, έχει κάνει μια συμμαχία με άλλους χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προετοιμάζουμε μια σειρά τροπολογιών και θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένες από αυτές. Προτείνουμε, για παράδειγμα, να ενισχυθεί η προστασία επενδυτή και καταναλωτή. Όλες οι εθνικές εποπτικές αρχές να έχουν στο καταστατικό τους ε, ως βασικό στόχο την προστασία του επενδυτή και του καταναλωτή. Προτείνουμε να ενισχυθεί η διοίκηση και η ανεξαρτησία των διοικητικών συμβουλίων της ΕΣΑ, η για να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ του χρηματοπιστωτικού κλάδου και των εμπειρογνωμόνων των ειδικών για τις πωλήσει λιανικής. Και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τα stakeholder groups. Στηρίζουμε τις προτάσεις για την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως, δυστυχώς, η πρόταση της Κομισιόν αποκλεί αντίστοιχο επίπεδο προστασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες που επενδύουν άμεσα στην οικονομία, όπως είναι οι ε, ατομικοί επενδυτές. Και θέλουμε ένα νέο ε, σύστημα συλλογικών αποζημιώσεων που να καλύπτει τους ατομικούς ε, μικροεπενδυτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναφέρει την εμπιστοσύνη του κοινού στην αγορά των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Εγώ είμαι από τη Γερμανία και έχω με εξετάσει όλη την περίπτωση της Volkswagen με χιλιάδες επενδυτές, με χιλιάδες και εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που παραπλανήθηκαν. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτό. Μας δείχνει πόσο χρειάζεται ένα σύστημα συλλογικών αποζημιώσεων για να αποζημιωθούν οι επενδυτές αυτοί που παραπλανήθηκαν και παραπληροφορήθηκαν. Δύσκολα θα επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Δύσκολα θα τους επαναφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Κεφάλαια Αγορά και Κεφαλαιακή Ένωση χωρίς να υπάρχει τέτοιο σύστημα συλλογικών αποζημιώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Τίμωθη Σάκεσμπη, εμπειρογνώμονας είναι ο, επό... ο επόμενος ομιλητής. Είναι η Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσω σήμερα ε, για να σας δώσω την ε, άποψή μου ε, του θέματος όσον από την πλευρά των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων ένα μεγάλο μέρος των ε, προγραμμάτων αποταμίευσης αφορούν ακριβώς αυτά τα προϊόντα. Ε, πρέπει να πω ότι για μας πάντα οι καταχρηστικές ε, πωλήσει ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι οι πρόσφατες ρυθμίσεις και νομοθεσίες οπωσδήποτε θα φέρουν κάποιες αλλαγές. Τρίτον, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αισθίωση όσον αφορά την επιτήρηση και περιορισμό των πρακτικών και τέλος θα δώσω και και κάποιε πληροφορίε κάποια στοιχεία όσον αφορά τι μελλοντικέ προοπτικέ. Ε, καταχρηστικές πωλήσει πρώτα απ' όλα. Ε, θα ήθελα να πω τρία πράγματα ε, όσον αφορά τα όσα έχουμε μάθει και από τα όσα βλέπουμε. Οι καταναλωτέ προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν τι σημαίνουν ακριβώς αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Χρειάζονται παιδαγωγία λοιπόν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει η συμπεριφορά των αγοραστών και των καταναλωτών να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Δεύτερον, όσον αφορά τις συγκρούσεις ε, συμφερόντων, καθώς επίσης ε, και τις προσωπικές κινητροδίες όσον αφορά την προστασία τέτοιων προϊόντων. Ε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι συγκρούσεις δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα και βεβαίως εμείς προσπαθούμε να τις διερευνήσουμε. Τρίτον, η υπερπλοκότητα των προϊόντων εξακολουθεί να είναι πρόβλημα. Ας πούμε, η δυνατότητα ας πούμε κάποιων προϊόντων που δίνονται ως επιβράβευση και τα οποία δεν εξηγούνται ακριβώς οι κίνδυνοι μπορεί να είναι κάτι ε, πάρα πολύ σημαντικό. Στο EBBI ε, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία αυτά αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει περισσότερο να ληφθεί υπόψη ε, το, να ληφθούν υπόψη οι συγκρούσεις. Τα σκάνδαλα δεν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται στην συνήθη πραγματικότητα. Δεύτερον, το θέμα της νομοθεσία ναι, βεβαίω θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ναι, την σωστή διακυβέρνηση, την ε, διαφάνεια κλπ. Βεβαίως ακόμα δεν έχω έχουμε γνώση και εμπειρία για το τι λειτουργεί σωστά ή τι δεν λειτουργεί για την ώρα. Ας πούμε, πολύ συχνά αναφέρεται ότι η συμμόρφωση τύπου tick box δεν ε, διασφαλίζει την ε, ε, σωστή αντιμετώπιση των καταναλωτών. Κατά αυτή την έννοια, το BIFID και το IDD είναι πολύ μεγάλα βήματα προς τα εμπρόσω και δημιουργούν πολύ νέε προσδοκίε όσον αφορά την επίλυση των θεμάτων υπέρ ε, του συμφέροντος των ε, καταναλωτών. Εμείς ε, η ΑΙΟΠΑ δουλεύουμε σκληρά έτσι ώστε οι καλές αρχές οι οποίες ενδεχομένως περιλαμβάνονται να ενδυναμωθούν και επομένως να μπουν κατά κάποιο τρόπο στην ζωή. Τρίτον, η επιτήρηση. Χρειάζεται οπωσδήποτε καλύτερη επιτήρηση γιατί αυτή δεν είναι ακόμα η ικανοποιητικοί. Οι πόροι οι οποίοι δίνονται ε, στην διαδικασία αυτή δεν είναι ικανοποιητικοί και πρέπει οπωσδήποτε καλύτερα να κατανοήσουμε ε, τις ε, συνθήκες και τους όρους του παιχνιδιού. Κατά την έννοια αυτή εμείς δουλεύουμε με τις NCAs έτσι ώστε να δώσουμε κάποιες ε, καλύτερες ε, δυνατότητες. Επίσης ε, δουλεύουμε για τα big data καθώς επίσης και για τις ταξιδιωτικές ασφαλίσεις. Προχωρούμε σε καλύτερη ανάλυση προϊόντων. Έχουμε επίσης ένα πρόγραμμα επίσκεψης των εθνικών αρχών επιτήρησης και τέλος συνεργαζόμαστε και με πλατφόρμες έτσι ώστε να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις σε προβλήματα διασυνοριακά. Πιστεύουμε ότι μέσω συνεργασιών τέτοιου είδους μπορούμε να, κάνουμε ε, καλές ε, πρακτικές, να έχουμε καλές πρακτικές. Ε, τέλος, να πω δύο λόγια όσον αφορά τις καινοτομίες. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προκύψουν κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις και όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά σχήματα και όσον αφορά τα ασφαλιστικά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε πώς εκεί που έχουμε καταχρηστικές πωλήσει μπορούμε να μετατρέψουμε, να αντιστρέψουμε την την ε, κατάσταση. Θα πρέπει να είμαστε, ε, ε, να κινούμαστε με τρόπο προληπτικό, με τρόπο προενεργητικό, έτσι ώστε να αποφύγουμε καταχρηστικές πωλήσει, όχι μόνο έτσι όπως τις βλέπαμε στο παρελθόν, αλλά έτσι όπως διαγράφονται και για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ιτμαν Λούντερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επικεφαλής του, του Τμήματος Αξιογράφων. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που δίνετε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει μερικά λόγια. Είναι πολύ δύσκολο να ακολουθεί κανεί τον κύριο Σέξπιρ που, ήταν, που ήταν και ειδικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν πολύ εύστοχε ε, οι παρατηρήσει του. Φοβούμαι ότι εγώ θα υστερήσω ε, συγκρινόμενος μαζί του, αλλά έχω και εγώ μια δομή. Θα μιλήσω πρώτα λοιπόν για το τι αλλάζει η ΜΥΦΙΤ 2 σε σχέση με την υπαριθμόν 1, γιατί τώρα από τα σκάνδαλα που αναφέρονται στην εξαίρετη έκθεση που έχει αναθέσει το Κοινοβούλιο να εκπονηθεί, αφορούν την περίοδο 2008-2012. Ε, πριν από την θέση εφαρμογή του 2018 της ε, νέας ε, νομοθεσίας MIFID 2. Επομένως, θα σας εξηγήσω τι βελτιώνει η νομοθεσία αυτή. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στα κενά του, τα ενδεχόμενα κενά στο ρυθμιστικό πλαίσιο και επίσης με βάση τα όσα είπε και ο Τίμωθη πάνω στην ίδια γραμμή λίγο πολύ, ε, θα αναφερθώ και σε ζητήματα υλοποίηση και την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας τελικά. Μη 2 πρώτα. Εδώ βελτιώνονται κάποια στοιχεία που οδηγούσαν, κάποια ε, σημεία που οδηγούσαν σε καταχρηστικές ε, πωλήσει. Παραδείγματι, εδώ έχουμε υποχρεωτική αποκάλυψη στοιχείων ε, μια σειρά κινδύνων που προηγουμένως δεν είχαν τονιστεί. Και έτσι έχουμε αυτήν την αλλαγή σε σχέση με, την περίοδο που με τα όσα ίσχυαν πριν την περίοδο 2018 ενημέρωση για κίνδυνο bail-in, δηλαδή υποχρέωση συμμετοχής στο κίνδυνο, ε, κίνδυνο σχετικό με ε, παράγωγο χρέος, με δευτερογενές μάλλον χρέος, κίνδυνο αφαιρεγγιότητας, ε, κίνδυνο σχετικό με τις αγορές στόχων, γιατί εδώ το θέμα δεν είναι να ο ε, πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται το προϊόν, αλλά και τα λοιπά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η αγορά και ο πληθυσμός ε, στον οποίο απευθύνεται προς πώληση το προϊόν. Το δεύτερο δευτερογενέ χρέο, ε, οι μετατρέψιμε αξίε, όλα αυτά απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό και πρέπει να περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του. Μια σειρά από προϊόντα βγαίνουν από το χαρακτηρισμό των μη περίπλοκων προϊόντων που μπορούν ε, να ε, πολλούνται στο σημείο πώληση χωρίς περαιτέρω εξηγήσει. Όλα τώρα περιγράφονται ω περίπλοκα και κυρίως αυτά που είχαν βρεθεί και στη ρίζα των προβλημάτων, ε, οι μεταβλητές, οι μετατρέψιμες αξίες ε, και άλλα στοιχεία που είχαν να κάνουν με τον πελάτη Λιανικής. Αυτά δηλαδή ήταν στη ρίζα των προβλημάτων που επεσήμανε και η έκθεση του Κοινοβουλίου εδώ λοιπόν πάλι έχουμε τα χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου, τον έλεγχο σε εθνικό ή αν υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ε, δραστηριοτήτων πολίτσεων, Βεβαίως πολλές είναι αυτές οι βελτιώσεις που επισημαίνουμε. Ε, βελτιώνεται πολύ η κατάσταση. Δεν είμαστε μία σχέση βέβαια στο σημείο που το 2008-2009, εκεί που είδαμε αυτά τα τόσο θλιβερά και λυπηρά γεγονότα. Αλλά αν μπορώ να το πω έτσι, το κύριο ζήτημα που δεν έχουμε αντιμετωπίσει είναι αυτό το οποίο έχει το Κοινοβούλιο σοφά ε, επισημάνει ως προβολή ιδίου χρέους. Δηλαδή, προβάλλεται το ίδιον χρέος, καλούνται και οι εργαζόμενοι να ε, επενδύσουν σε αυτό κτλ. Επομένως, εδώ μπορεί να υπάρχει ένας στόχος πώληση μέρους του χρέους προς τον ε, πελάτη της Λιανικής, αφενός, αφετέρου όμως υπάρχει και η πρόκληση να εξηγήσει κανείς γιατί είναι πρόσφορο για τον ιδιώτη επενδυτή το εν λόγω χρέος. Επομένως, ένας ταξιούχος που κάθεται στο τραπέζι ε, και του εξηγούμε ότι πρέπει να πάρει ε, να κάνει επένδυση πάνω στο σταξιοδοτικό προϊόν. Προφανώς υπάρχει ε, στο σταξιοδοτικό προϊόν της εταιρείας στην οποία εγώ δουλεύω που θέλω να το πουλήσω, προφανώς έχω σύγκρουση συμφερόντων, γιατί θέλω να πουλήσω και μου έχει πει και ο εργοδότη μου ότι πρέπει να πουλήσω, αλλά σε εκείνον ίσω να μην είναι το ίδιο συμφερόν. Επομένω, εδώ είναι ένα κενό της νομοθεσίας, η σύγκρουση συμφερόντων που πρέπει να αποφεύγετε πρέπει να αντιμετωπίσετε. Ωστόσο αναφέρεται σε ένα άρθρο ότι εάν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή δεν μπορεί να περιοριστεί η σύγκρουση συμφερόντων, τότε πρέπει να αποφεύγει την πώληση ο ε, πολιτής του συγκεκριμένου προϊόντος. Μα εδώ ακριβώς είναι η κατάφορη παραβίαση αυτής της υπορήτρας που βλέπουμε ότι ο πολιτής δεν αποφεύγει, δεν ε, προχωρεί σε αποχή από την πώληση των εν λόγω αξιών που ε, ε, είτε έχουν μεγάλο κίνδυνο, είτε εν πάση περιπτώσει εκπροσωπούν μια σημαντική ε, σύγκρουση συμφερόντων. Εδώ λοιπόν υπάρχει το κενό, αυτό πρέπει να καλυφθεί από πρόσθετη νομοθεσία. Έχουμε εξηγήσει ότι η σύγκρουση συμφερόντων πρέπει πάντα να αποφεύγεται. Και καταλήγω στο ότι πολύ μεγάλο κομμάτι της νομοθεσίας έχει ολοκληρωθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το big selling είναι παραδείγματι, περίπλοκο θέμα, αλλά όπως είπε και ο Τίμωθη πριν από μένα, η έμφαση τώρα πια πρέπει να έρθει στην συγκεκριμένη εφαρμογή, στο εγχειρίδιο, στο σημείο πώληση και εκεί ακριβώς ξέρουμε πολύ καλά ότι με το σύστημα του ΣΥΛΟ της δέσμης πολλούνται μια σειρά προϊόντων. Επί παράδειγμα, θέλει κανεί να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, η τράπεζα του λέει και πολλέ φορέ και υποχρεωτικά ότι κοίταξε πρέπει να πάρει αυτή την ασφάλιση γιατί έχουμε την ε, ε ομαδική ασφάλιση για να πάρει ένα καλύτερο επιτόκιο στο κτηματικό σου δάνειο και το καθεξής. Έρχεται λοιπόν και τον πιέζει με το σύστημα του ΣΥΛΟ να πάρει και άλλα προϊόντα. Αυτό δεν έπρεπε να επιτρέπεται. Είναι απλά τα πράγματα γιατί υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, υπάρχουν εσωτερικά προϊόντα τα οποία δεν είναι απαραίτητα καλύτερα και δεν πρέπει να προτιμούνται από αυτά των ε, ανεξαρτήτων ε, ανταγωνιστών. Αυτό θα αλλάξει όχι μόνο με ένα εγχειρίδιο, αλλά οπωσδήποτε με αλλαγή νοοτροπίας. Δεν πρέπει να έχει ανταπόδοση για τον εργαζόμενο η δυνατότητα πώληση μια σειρά από προϊόντα ως το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού, αλλά η ικανοποίηση του πελάτη, το καλύτερο προϊόν που θα πωλήσει τον πελάτη. Πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε και συμφωνώ με τον Τίμωθη η ευαισθητοποίηση, η παιδαγωγική δουλειά που θα γίνει, αλλά και η αλλαγή της θέσης της κοινή γνώμη που θα πρέπει να διεκδικήσει καλές και ανεξάρτητες συμβουλές. Ακόμα και αν το προϊόν του το πουλάει μια τράπεζα. Uh, Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές για την εξαιρετική τους παρέμβαση, την τρομερά χρήσιμη. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής μας. Παρακαλώ ζητήστε το λόγο όσοι ενδιαφέρεστε να τοποθετηθείτε. Ο κύριος Ουρτασόν, παρακαλώ. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα τα ισπανικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας, πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και έχουμε οργανώσει αυτή την ακρόαση λόγω του μεγάλου αριθμού των αναφορών Ευρωπαίων πολιτών που έπεσαν θύματα καταχρηστικών πωλήσεων και εξετάζουμε αυτά τα πράγματα για να δούμε ποια ε, νομοθετική, ποιες αλλαγές πρέπει να επιφέρουμε στη νομοθεσία για να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές καταχρήσεις τα τελευταία χρόνια σε όλα τα είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων, στα ενυπόθηκα δάνεια, έχει γίνει χαμός γενικά. Είναι εξαιρετικές οι εκθέσεις και μας ενημερώνουν ιδιαιτέρως, μας διαφωτίζουν πολύ για το ποιες νομοθετικές αλλαγές πρέπει να επιφέρουμε. Θα ήθελα να θέσω ορισμένες ερωτήσεις στον παρεμβαίνοντες. Πρώτα στον κύριο Λούντερ, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή του. Μιλήσατε για τις κατεξουσιοδότησες πράξεις για το self-placement. Αυτό που περιλαμβάνει η κατεξουσιοδότηση πράξη αρκεί. Δεν το ξέρω αυτό, δεν είμαι βέβαιο γιατί στην τελευταία φράση για τη σύγκρουση συμφερόντων λέει «may refrain», δύναται να απόσχει. Δεν είναι αρκετά ισχυρή αυτή η διατύπωση για να ε, προληφθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη διατύπωση, έτσι δεν είναι. Ποια είναι η άποψη σας από αυτό. Δεύτερο ερώτημα για το BRRD, για την οδηγία για την εξυγίαση των τραπεζών και την ε, ε, ε, διάλυση αυτών και την εκαθάριση αυτών. Bank Recovery και Resolution Directive. Εδώ τίθεται δύο θέματα. Δηλαδή, όταν ε, κλείνει μια τράπεζα και εξηγένεται, υπάρχουν προϊόντα που έχουν πολιθεί με παράνομο τρόπο. Τι κάνουμε με αυτά. Τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ειδικά κεφάλαια για την αποζημίωση. Αυτό ήταν η Ιταλική περίπτωση. Έχουμε σύστημα εγγύηση καταθέσεων, έχουμε το Ταμείο Εξυγεύσης Τραπεζών. Άλλη επιλογή προτείνεται από την έκθεση είναι να απαγορευτεί εξ αρχής να εφαρμόσετε το bail-in σε αυτούς που διακρατούν προϊόντα τα οποία έχουν πολιθεί με ε, παράνομο τρόπο. Να μην υποχρεούνται δηλαδή να συμβάλλουν οι ίδιοι στη διάσωση και εξοικίαση της τράπεζας από τη στιγμή που αγόρασαν προϊόντα που τους είχαν πολιθεί κακόπιστα και καταχρηστικά. Ποια είναι η άποψή σας ε, για τις δύο αυτές επιλογές. Και τέλος, Ρομπέρτο, Άλλο σημαντικό θέμα είναι οι κυρώσεις. Π.χ. στα ενυπόθηκα δάνεια και σε αυτά που έχουν γίνει. Στην ισπανική περίπτωση, για παράδειγμα, η Τράπεζα της Ισπανίας έχει βούληση να μην αναλάβει δράση και να μην τιμωρήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ουσιαστικά είχαν πωλήσει ενυπόθηκα δάνεια με ε, ε, δόλιο ή τέλο πάντων νομικός μαχητό τρόπο. Θα ήθελα την άποψή σας επ' αυτό. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ε, εν τω μεταξύ, μέχρι να αποφασίσουν οι συνάδελφοι να θέσουν ερωτήσεις, να δώσω το λόγο στους ε, απαντώντες, να πω εγώ κάτι εν τω μεταξύ. Ε, σε συνέχεια της ερώτησης του κυρίου Ορτασούν και απευθύνομαι σε όλους τους ε, ομιλητές γιατί έχουμε διατυπώσει με πολύ μεγάλη προσοχή και έχουμε διαβάσει με πολύ μεγάλη προσοχή τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και τη δήλωση της Ευρωπαϊκής, Τραζι... Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για τη διακράτηση τίτλων ε, και για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και για όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο και φαίνεται αυτό ξεκάθαρα από τις δηλώσεις αυτές, να έχουμε μία απλή λύση γιατί κανείς βεβαίως δεν θέλει να πει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να υπαχθεί σε μπέιλιν, γιατί αν δεν μπορεί να υπαχθεί σε μπέιλιν δεν μπορεί και να απολυθεί. Αν απολυθεί σωστά, τότε ο επενδυτής που το αγοράζει αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Άρα, αφού θέλει υψηλότερη απόδοση, γιατί να πρέπει να αποζημιωθεί και να μην μπει στο μπέιλιν. Είναι πολύ λογικό. Από την άλλη δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα που να λέει ότι αυτά τα προϊόντα θα αποκλείονται εξ αρχής. Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις καταχρηστικών πωλήσεων. Έχουμε ένα ολόκληρο απόθεμα τέτοιου είδους χρηματοπιστωτικών προϊόντων που πωλήθηκαν καταχρηστικά. Τίθεται το ζήτημα της αποζημίωσης. Μετά έχουμε το θέμα της ροής, η οποία βαίνει μειούμενη όμως η τάση είναι καθοδική, όμως πώς τη βλέπετε εσείς. Πάμε πράγματι προς την εφαρμογή και υλοποίηση των νέων κανόνων. Που δημιουργούν ε, ένα επίπεδο καταχρηστικών πωλήσεων πολύ μικρό και άρα βιώσιμο. Ή νομίζετε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι εκτός από όλα αυτά που έχουμε κληρονομήσει καταχρηστικές πωλήσει προϊόντων του παρελθόντος και τι κάνουμε με αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, υπάρχει και ροή δημιουργίας νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων που δύναται να απολυθούν καταχρηστικά. Ήταν πολύ καλή η δήλωση των δύο ευρωπαϊκών αρχών όμως εκεί αναδεικνύουν το ενδεχόμενο μιας αντίφασης μεταξύ των δύο φαινομένων. Επομένως, παίρνω τη σκητέλα από τον κύριο Ουρτασούν για να σας ζητήσω να τοποθετηθείτε σε περισσότερο βάθος ως προς αυτά τα ζητήματα. Ο Σβέν Κίγκολντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας... Και ευχαριστώ ιδιαιτέρως για όλες αυτές τις μελέτες, για την ενημέρωση που μας προσφέρατε και σήμερα. Και βέβαια σε όλη τη δικασία κάποια από εσάς. Θα επισημάνω ένα-δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, και απευθύνομαι στην Επιτροπή, στις ε, μελέτες αλλά και στην παρουσίαση σήμερα και στα δημοσιεύματα που αναφέρονται για την ε, καλύτερη, για το Better Finance σήμερα, βλέπουμε σημαντικές παραβιάσεις ή μη τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Και έτσι ρωτώ το Τίμαν Λούτερς. Τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε από εδώ και μπρο. Έτσι ώστε να εφαρμόζεται αποτελεσματικά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όπως αναμένει ο πολίτης. Στους συγκεκριμένους τομείς. Στο κλειστό δίκτυ, το self-placement, όλα αυτά που αναφέρατε εσείς δηλαδή πώληση ιδιών προϊόντων, πιθανές ε, παραβιάσεις της MCD που αναφέρονται οι μελέτες. Μπορείτε λοιπόν εσείς να δεσμευτείτε ότι θα παρακολουθείτε στενά όλη αυτή την τήρηση της δουλειάς που έχουμε κάνει για να υπάρχει υψηλό επίπεδο σεβασμού στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Για την ΑΕΟΠΑ, η επόμενη ερώτηση. Διάφοροι παράγοντες στην αγορά μου μίλησαν για κάποια ζητήματα ε, προβλημάτων στην ασφάλιση πληρωμής χρέους. Όπως για παράδειγμα τον αγοράζει κανείς ένα αυτοκίνητο που του πουλάνε μαζί πακέτο ή το ίδιο και στην αγορά ενός ε, ε, ταξιδιού. Α, Ιταλία, α πούμε, μα αρέσει πολύ να πηγαίνουμε στην Ιταλία, άσχετο αν θα μα καταγράφουν σε κατα, κάποιο παράξενο ε, τρόπο. Κατά την κράτηση λοιπόν του ε, εισιτηρίου προσφέρεται και ένα προϊόν ασφάλισης. Γενικά, προστασία πώληση. Το ίδιο και στην αυτοκινητοβιομηχανία, δηλαδή στη Γερμανία. Ξέρω ότι η προμήθεια του πολιτή της ε, αντιπροσωπείας εξαρτάται και από το αν θα πωλήσει ε, αυτή την ασφάλεια πληρωμής στον αγοραστή και μάλιστα η προμήθειά του μπορεί να πάει μέχρι και το 70% αυτής της ασφάλειας. Ερωτώ λοιπόν την ΑΙΟΠΑ. Αυτές τις εμπορικές πρακτικές τις έχετε κοιτάξει. Και αν όχι, είστε διατεθειμένοι να ξεκινήσετε μια σοβαρή διερεύνηση, εξέταση αυτών των κατάφορων παραβάσεων των αρχών του δικαίου που εκδηλώνονται σε αυτή την αγορά. Επίσης, εδώ έχουμε να κάνουμε με καταχρηστικούς τόκους υπερβολικά υψηλούς, ε, με καταχρηστική μάλλον ε, συνθήκη σε σχέση με, την, ε, με το υπερβολικά υψηλό κόστος σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται. Για την ΑΙΟ πάλι μια ερώτηση για, την καλύτερη, για το Better Finance. Ε, πώς βλέπετε να προχωρά σε σχέση με τις πιο πρόσφατες αλλά και τις παλαιότερες εμπειρίες σας. Ήταν ικανοποιητική η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν ε, τη συγκρίνουμε με τα ε, προβλήματα που είχαν εντοπιστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου. Για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ εκ μέρους ομάδας μου όλους ομιλητές. Θα, θα, θα κοιτάξω να δοθεί και συνέχεια. Λυπούμε βαθύτατα σημειώνω κοιτώντα γύρω μου ότι, για το γεγονό ότι μόνο δύο πολιτικέ ομάδε εκπροσωπούνται εδώ, ενώ η κεντροδεξιά του Κοινοβουλίου φαίνεται πω δεν θεωρεί αυτά τα θέματα ιδιαίτερη προτεραιότητα. Βλέπω βεβαίω του συμβούλου των ομάδων και του ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ. Αλλά νομίζω ότι ο χρηματοπιστωτικός καταναλωτής χρειάζεται και αξίζει περισσότερο σεβασμό από το Κοινοβούλιο. Συμμερίζομαι και εγώ τις παρατηρήσεις του Σβέν και καλώ τους ομιλητές μας να ξεκινήσουν. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Ποιος θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τα δύο επιπλέον ζητήματα τα οποία έρθισαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, η διατύπωση που έχουμε εισαγάγει είναι πιο αυστηρή λίγο πιο αυστηρή. Δεν λέει εάν δεν έχετε, εάν έχετε ε, ενδεχομένω θα αποτρέψετε, λέει ότι αν έχετε τέτοιου είδους δυσεπίλητα, ε, τότε θα πρέπει να λάβετε ε, υπόψη την δυνατότητα you shall refrain from. Επομένως, από τη στιγμή που υπάρχει διαπιστωμένη σύγκρουση συμφερόντων, τότε ε, θα λάβετε τα μέτρα σας έτσι ώστε... Εάν, εάν ε, στην πράξη, στην ε, αντιμετωπιστεί με τον τρόπο αυτό από το σημείο πώληση, τότε υπάρχει ζήτημα. και έρχομαι στο ερώτημα του Σβεν Κίγκολτ. Ε, κάποια στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε λίγο στον πραγματικό κόσμο, να φύγουμε από το ε, προστατευμένο έτσι, περίβλημά μας και να πάμε ε, στον κόσμο να μιλήσουμε, να μιλήσουμε στους τριμερείς διαλόγους γιατί πολλά κάνουμε μεταξύ μας αλλά δεν βγαίνουμε προς τα έξω στα διάφορα φόρα των εμπλεκομένων πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουμε σε ε, εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ε, είναι πολύ καλό ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχετε έτσι καλή εμπειρία όσον αφορά τέτοιες περιπτώσεις να βγαίνετε προς τα έξω και να μιλάτε εμείς. Θα έχουμε και κάποια εκδήλωση που θα αφορά το MIFID έτσι ώστε να εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνουν οι κανόνες, περί τίνος πρόκειται και επομένως να αυξηθεί η επίγνωση των πραγμάτων αυτών και των θεμάτων αυτών. Επίσης υπάρχουν οι μόνιμε επιτροπές ΕΣΜΑ, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε στην μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών να ε, συζητιούνται καθημερινά τα πράγματα. Ξέρετε, αυτή είναι καθημερινός αγώνας που πρέπει να δώσουμε, να μιλάμε με τους ρυθμιστές, να μιλάμε με τις ρυθμιστικές, ε, ρυθμιστικές αρχές, με σαφήνεια και το ζήτημα των σημείων πώληση θα πρέπει να καταλάβετε ότι το θέμα τα μία πώληση είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελέγχεται κεντρικά από τις Βρυξέλλες γιατί συμβαίνει ε, σε δεκάδες χιλιάδες ε, ε, συζητήσεις. Θα πρέπει, ναι, είναι γεγονός ότι όταν λαμβάνουμε γνώση θεμάτων τα αντιμετωπίζουμε. Οι σύμβουλοι οπωσδήποτε θα πρέπει να αναφέρονται στις ανάγκες των επενδυτών και οι εκπρόσωποι των επενδυτών θα πρέπει να μιλούν για τις ανάγκες των επενδυτών αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν γίνεται μονάχα με ανταλλαγέ εγγράφων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εργαλείο που λέγεται MIFID και ε, ε, οπωσδήποτε δεν αρκεί το να λέμε υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε και να το, ε, να το υπογράψετε στο τέλος. Ε, θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Οι νοοτροπίες αλλάζουν σιγά σιγά με περισσότερη εκπαίδευση, με περισσότερη παιδαγωγική ε, προσπάθεια και θα πρέπει οπωσδήποτε να δεσμευτούμε περισσότερο, να μάθουμε, να βλέπουμε τι γίνεται επί τόπου. Ίσως θα πρέπει να γίνουν και περισσότερες μελέτες. Έχουμε μια μελέτη για το follow-up του MIF Ενδεχομένω ενδεχομένως θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε κι άλλε μελέτε σχετικά με το τι συμβαίνει επί τόπου. Πρέπει να κάνουμε μελέτε, επιθεωρήσεις, έρευνε, mystery shopping επίση. Ε, ε, ε, Αυτέ οι διαδικασίε θα πρέπει να προωθηθούν έτσι ώστε να ξέρουμε τι συμβαίνει επί τόπου. Και επίση πιο σημαντικό ακόμα, αυτοί οι οποίοι δρούν επί τόπου να ξέρουν ότι κάποιο θα παρακούσει, κάποιο θα παρατηρήσει τι γίνεται στη διάρκεια αυτών των συζητήσεων και ότι ότι δεν πρόκειται πλέον για ανώνυμες μυστικές διμερείς συνομιλίες. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Προσυπογράφω αυτά που είπε ο προελίσσες ε, ε, σχετικά με το δεύτερο σκέλος και όσον αφορά ε, τον, το, το πρόβλημα το οποίο έγκυται στο πώς ε, οι κανονισμοί οι οποίοι υπάρχουν και οι κανόνες οι οποίοι υφίστανται θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κανονικά στην πράξη ε, στις μεγάλες, στις μεγάλες τράπεζες, πώς λαμβάνουν χώρα οι συζητήσεις, τα ζητήματα προστασίας τα οποία προκύπτουν Γι' αυτό πραγματικά θα πρέπει η επιτήρηση, θα πρέπει η ε, σωστή εφαρμογή να αποτελέσουν τα σημεία ε, εστίασής μας. Αυτό το γνωρίζουμε, έχουμε επίγνωση ε, των θεμάτων αυτών. Είχαμε μεγάλες αλλαγές όμως τα τελευταία χρόνια ε, στους κανονισμούς και προσπαθούμε με πρακτικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε όλες τις αλλαγές αυτές. Επομένως, απολύτως προσυπογράφω. Το mystery shopping, κοιτάξτε, εμείς το κάναμε αυτό και είδαμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στη, στα σημεία πώληση, όποιοι και αν είναι οι κανόνες, όποιοι και αν είναι οι κανονισμοί. Πραγματικά θα πρέπει αυτό το θέμα που αποτελεί μεγάλη πρόκληση να το αντιμετωπίσουμε με μεγάλη προσοχή. Ε, όσον αφορά το ε, θέμα του PPI γενικότερα, είναι ε, κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, το κατανοούμε, έχουμε συνείδηση του θέματος. Ε, έχουμε δουλέψει με καταναλωτές για πολλά χρόνια, έχουμε δουλέψει για το PPI ε, όσον αφορά τα σκάνδαλα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε και μάλιστα πρόσφατα αυτή την εβδομάδα συζήτηση με την Εθνική ε, Αρχή Επιτήρησης γιατί ξέρουμε ότι είχαν προβλήματα και ιδιαίτερους προβληματισμούς σε διάφορες αγορές. Πρόκειται οπωσδήποτε κάτι το οποίο παρακολουθούμε προσεκτικά. Ε, σας ανέφερα ότι κάνουμε έρευνα όσον αφορά τις ε, ταξιδιωτικές ασφαλίσεις, ε, ε, γιατί μπορεί να μην είναι υψηλής αξίας προϊόντα, αλλά πολλές φορές έχουν υψηλή προμήθεια. Αυτό δεν αποβαίνει πάντα προς ζημία του καταναλωτή, δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την διαχείριση ε, λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι ποτέ συμφέρουσα για το καταναλωτή αυτέ οι προτινόμενε ταξιδιωτικέ ασφάλειε, αλλά ε, διατρέχει, υπάρχει πάντα ο κίνδυνο υπερασφάλιση άνευ λόγου. Εμεί παρακολουθούμε λοιπόν τα θέματα αυτά. Αυτό το κάνουμε ήδη άλλωστε και ε, αποστάλουμε ερωτηματολόγιο σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ε, του κλάδου ε, και στο τέλος του καλοκαιριού θα ε, βγάλουμε τα συμπεράσματά μας έτσι ώστε ενδεχομένως να ανεληφθεί δράση από το φθινόπωρο και μετά. Πρόκειται για αρκετά προβληματικό θέμα. Να συνεχίσουμε. Θέλετε να κάνετε μια, follow, μια συμπληρωματική ερώτηση. Νομίζω καλύτερα λέει ο Πρόεδρος να ολοκληρωθεί ο γύρος των ομιλητών και μετά. Ο κύριος Φέλπ, ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι στο θέμα του self-placement για ορισμένα προϊόντα υψηλού κινδύνου και τον τρόπο που το αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ο τραπεζικός τομέας για να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια ή τα κεφάλαια που είναι επιλέξιμα για το TLAC, την ε, ικανότητα απορρόφησης ε, συνολικών απολειών ή για το MRL, τι ελάχιστε απαιτήσει για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες απώλειες. Έχουμε νέους κανόνες και νομίζω ότι ως Εθνική Αρχή αλλά και ως Ευρωπαϊκή Αρχή έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται αυτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κανείς τόπου να πάει να δει εάν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Και πρέπει να τιμωρήσουμε σε ορισμένες περιπτώσεις και να επιβάλλουμε κυρώσεις και να το γνωρίζουν αυτό για να τηρεί τη διαδικασία. Ω εποπτική αρχή, λοιπόν, έχουμε την ευθύνη να επιβάλλουμε την συμμόρφωση με την νομοθεσία. Ήθελα να πω ότι στη Γαλλία, σε σχέση με αυτή την προβληματική, είναι πάρα πολύ ε, ε, σημαντικός ο τομέας των mutual, των αμοιβαίων ασφαλίσεων και των, και των αντασφαλίσεων. Άρα υπάρχουν καλές πρακτικές και άλλοι ασφαλίσεων τα mutual και υπάρχουν οροφές που επιβάλλονται και κατώτατα όρια επίσης για τους ε, για το υπαγόμενο ή δευτερεύον χρέος, για τους υπαγόμενου ή δευτερεύοντες χρεωστικού τίτλους, έτσι ώστε κανεί να μην έχει μια τρομερά ισχυρή έκθεση σε προϊόντα τύπου ιδίων κεφαλαίων από τη μία και από την άλλη πλευρά να μην ε, υπάρχουν ε, τέτοιου είδους δευτερεύοντε χρεωστικοί τίτλοι που μπορούν να επιφέρουν τέτοιου είδου εξελίξεις. Έχουμε δηλαδή οροφές και κατόφλια ε, που είναι πολύ σημαντικά και αυτά εννοούσα όταν μιλούσα για τις δυνατότητες επαναφοράς ε, διατυπώσεων για το ελάχιστο επίπεδο της ονομαστικής αξίας των τίτλων. Πρέπει αυτά να τα ε, συμπεριλάβουμε στην οδηγία για την εξυγίαση διάσωση ε, τραπεζών. Άρα ο εποπτικός μας ρόλος είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικός. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Θα ήθελα, λέει η κυρία Μπένερα από το Better Finance, να μιλήσω για το ερώτημα του ε, Σβέν Κίκολτ. Πράγματι, θεωρώ ότι πολύ περισσότερα θα, μπορούσαν, θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό συνεχώς ασκούμε πιέσεις για να επέλθουν αλλαγές. Και αν δω τα Key Information Document και το PRIP, η Χρειάζεται πράγματι αυτός ο στόχος αναθεώρησης του κανονισμού φέτος, αλλά δεν ελπίζω να συμβούν και πολλές καταιγιστικές εξελίξεις εντός του 2018. Αυτό θα περιμέναμε όμως να γίνει. Υπάρχει πολύ μεγάλη ασυνέπεια μεταξύ των κανόνων προστασίας των επενδυτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Έχουμε ε, το MIFID 2, το IDD, το PRIP, δηλαδή τα κανονισμό για ε, τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται στην ασφάλιση και πολλούνται προϊόντα λιανικής. Υπάρχουν πολλές αποκλήσεις λοιπόν στο επίπεδο προστασίας, άρα και η Επιτροπή και οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για να ενισχύσουν την εποπτεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Κύριος Μποντζοβάνη, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να απηχήσω κάποια από τα θέματα που υπενθύμισε ο κύριος Τσίλμαν. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έχει κάνει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το άρθρο 41 στο επεδοδίο και τις ειδικέ ε, μνήες στην αυτοπροβολή ή προβολή ιδίων προϊόντων. Πρέπει να υπάρχει νομοθεσία κάποια διάταξη η οποία να εξασφαλίζει ουσιαστική και αυστηρή εποπτεία στην περίπτωση προβολής ιδίων προϊόντων. Και επίσης, κάτι το οποίο ανέφερα και στην εισαγωγική μου παρατήρηση, θα επισημάνω ότι εμείς από το 2009 έχουμε προβεί σε ανακοινοθέντα το 9 και το 14 γιατί περίπλοκα, όπως ονομάζονται, προϊόντα. Και εκεί πάλι έχουμε την ε, μνήα των, της προβολής ιδιών προϊόντων από μεσολαβητές, από ενδιαμέσους. Η εμπειρία που έχουμε από το 2010 με 31% μειώνεται στο 10% το 2017 η προβολή ιδιών προϊόντων και άρα εάν υπάρχει διεθνής αλλά και εγχώρια νομοθεσία, εμείς ως αρχή αρμόδια μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα γιατί έχουμε αυτά τα εργαλεία στο χέρι μας. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή. Η άλλη που αντανακλάται και στις μελέτες σας, μελέτες που λάβατε, έχει να κάνει με την δυνατότητα για νομοθετική διαμεσολάβηση ή διαιτησία. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω τις διαφορές, τις τεράστιες διαφορές μεταξύ της θεωρίας και της ε, περιγραφής της ε, ε, προβολής ή της υποκίνησης σε αγορά ιδίων προϊόντων. Και εδώ θα υπενθυμίσω ότι η είναι μία ε, οδηγία και επίσης θα αναφέρω ότι υπάρχει ο ειδικό ε, κανόνας της IDD που έχει να κάνει με την υποκίνηση, αλλά έχει πολύ περιορισμένη ε, αυστηρότητα και εφαρμογή. Η IDD, η IDD λειτουργεί ως οδηγία ελάχιστης συμμόρφωσης ελάχιστων προδιαγραφών. Και αυτό σημαίνει σημαντικές δυσκολίες για τις αρμόδιες αρχές. Γιατί ο κλάδος, ο χρηματοπιστωτικός, αλλάζει σε ρυθμούς ταχύτητας από το ένα προϊόν ε, για να προβάλλει ένα άλλο. Εδώ όταν έχουμε να κάνουμε με επενδυτικά προϊόντα στηριζόμενα σε ασφαλιστική δραστηριότητα, και η κάλυψη των επενδυτικών με την, που στοχεύει η IDD, με την ελάχιστη κάλυψη ε, ως προς την υποκίνηση σε αγορά, είναι τόσο διαφορετικά τα προϊόντα αυτά που δεν μπορούν να καλύψουν τα ασφαλιστικά που θα πρέπει να καλύπτει η MIFID. Επομένως, αν δεν υπάρχει νομοθεσία δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Παρακαλώ, δεύτερη ερώτηση, παρακαλώ κύριε συνάδελφε. κύριος Γκίγκολτ για να αντιληφθώ περισσότερο, για να γίνει κατανοητό αυτό που κάνει η ΑΙΟΠΑ ή αυτό που δεν κάνει. Σε σχέση με την ε, ασφάλιση προστασίας πωλήσεων, έτσι, ε, μας λέτε ότι υπάρχουν ε, διάφορες λύσεις, μας είπατε εσείς για τα ταξίδια, εγώ αναφέρθηκα και στην, στα δάνεια, τα καταναλωτικά για αγορά αυτοκινήτου, μεγάλος τομέας, αφορά πολλούς καταναλωτές. Ε, το ίδιο στον το χρηματοπιστωτικό τομέα. Δηλαδή εσείς τώρα αυτούς τους τομείς τους καλύπτετε και ποια είναι τα μέτρα που ενδεχομένως συζητάτε στο πλαίσιο αυτής της ε, δουλειάς σας και πώς μπορείτε να βοηθήσετε το κοινό να αντιληφθεί καλύτερα το ποσοστό της προμήθειας που καλύπτεται μέσα σε αυτή, που ε, κρύβεται μέσα σε αυτή την αγορά απλό, μια απλή μεζούρα για να καταλάβει ο πελάτης εάν έχει αξία το προϊόν που του πουλάνε ή αν είναι σκέτη κερδοσκοπία. Και βεβαίως υπάρχουν προϊόντα στην αγορά που είναι χρήσιμα. Αλλά αν η ε, προμήθεια για την πώλησή τους ανέρχεται στο 70% νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. Και ασφαλώς η ΑΕΟΠΑ πρέπει να είναι πολύ πολύ αυστηρή ως προς την προστασία από την κερδοσκοπική εκμετάλλευση του καταναλωτή. Ποιες ε, αγορές καλύπτεται. Θέλω αυτό να είναι σαφές. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και οι περισσότεροι καταναλωτές νομίζω αν γνώριζαν τι συμβαίνει θα ήταν... Ε, θα αισθάνονταν βαθύτατη απογοήτευση. Ναι, παρακαλώ, έχετε να απαντήσετε. Κοιτάξτε, για να μπορούμε να διαχειριστούμε το θέμα, τη δουλειά όλη αυτή, τον όγκο της εργασίας, ε, σχολούμαστε τώρα με την ασφάλιση στα ταξίδια, αλλά πάλι ενδεικτικό είναι αυτό. Ας πούμε ότι είναι ένα είδος πειραματικής προσέγγισης, πιλωτικής προσέγγισης για να δούμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε και τις υπόλοιπες μορφές ε, τη ε, της ιδίων προϊόντων με την κατανομή και τα λοιπά, πώς λειτουργεί και σε επίπεδο επιτροπής, πώς μπορούμε να το αναλάβουμε, πώς μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, να κατανοούμε τη δουλειά, να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί η αγορά αυτά. αυτή. Η προμήθεια μπορεί να είναι και πάνω από 70% σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που μπορεί κανείς να αναπτύξει με τον κλάδο γύρω από την έννοια του αποδεκτού και μη ή προσήκοντος και μη επίπεδου προωθήσεις ιδιών προϊόντων. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε συμπεράσματα. Μάλλον δεν θα ε, είναι όμως συμπεράσματα που να λένε ότι πρέπει να απαγορεύεται η προβολή, η πώληση αντίστοιχα ασφαλιστικών προϊόντων. Αλλά κάποια όρια, κάποια ε, περιορισμοί και αυτό, όπως είπα, θα πρέπει να ανοίξει και σε άλλες αγορές για άλλα προϊόντα που και εσείς αναφέρατε. Ασφάλιση αποπληρωμής δανείου, επί παραδείγματι, πολύ ενδιαφέρουσα, με διαφορετικές μορφές σε διάφορες αγορές. Ε, μπορεί όμως τα θέματα να μην είναι τόσο διαφορετικά, οι συγκρούσεις συμφερόντων τόσο διαφορετικές. Εν πάση περιπτώσει ξεκινούμε από έναν τομέα, από ένα κλάδο συγκεκριμένο για να μπορέσουμε μετά να ανοιχτούμε και να καλύψουμε και τους υπόλοιπους. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η αναθεώρηση, θεματική αναθεώρηση τη λέμε, thematic review για φέτος, για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα και μετά να δούμε πού μας οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ξέρετε, έχουμε θέμα νομικού πλαισίου. Στα συμπεράσματα θα εντοπίζονται ίσως τομείς στους οποίους χρειάζεται κάποια περαιτέρω μελέτη ή ίσως κάποιοι άλλοι στους οποίους θα συμβουλεύουμε την νομοθετική παρέμβαση. Αυτά. Ωραία. Εσείς τουλάχιστον σημειώνετε εκ μέρους της δικής μας της ομάδας ότι εμείς θέλουμε το ταχύτερο δυνατό δράση και όχι να περιμένουμε με να τελειώσει ο χρόνος και να παραμένουμε απαθείς και αδρανείς ενώ ε, λαμβάνει η χώρα εκτεταμένη κερδοσκοπία. Η Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω, λέει η κυρία Περβάος Μπερές, γι' αυτό λοιπόν κάθομαι στο έδρανο του Προέδρου. Δεν έχω παρακολουθήσει την ανταλλαγή απόψεων, δεν ξέρω ακριβώ ποιο θέμα συζητείτε. Από τους... Στρέφομαι του παρεμβαίνοντε. Ε, θέλει κάποιο να απαντήσει τον συνάδελφο κύριο Σβεν Κίγκολτ. Α, έχει ήδη απαντηθεί το ερώτημα. Άμα θέλει μπορεί να επανέλθει ο κύριο ε, Κίγκολτ. Άρα, μπορώ να κηρύξω το πέρα στη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ θερμά. Από ό,τι καταλαβαίνω, ε, η συνεισφορά σας ήταν πολύ σημαντική για να προβληματιστούμε για τη συνέχεια που θα δώσουμε, ειδικά για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε την ε, αναθεώρηση της ESA και αν πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες παρέμβασης των ε, αρχών αυτών σε σχέση με αυτά τα προϊόντα θα το δούμε πολύ προσεκτικά. Υπάρχει και ένα θέμα με το PRIP, Package Retail Insurance Based Investment Product, με το, αυτό τον κανονισμό. Επομένως, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρουσία τους, για τη συμμετοχή τους, για τη συνεισφορά τους για την εξέταση αυτού του σημείου στην ημερήσια διάταξη, το οποίο το συμπεριλάβαμε στην ημερήσια διάταξή μας, γιατί έχουμε πάρα πολλές αναφορές σχετικά, σχετικές με το θέμα από Ευρωπαίους πολίτες που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή Αναφορών. Δεν πρέπει μόνο να ασχολούμαστε με τους κανονισμούς και τα μακροοικονομικά ζητήματα, αλλά και με αυτό αυτό το σκέλος ε, το πολύ πρακτικό και πολύ σημαντικό για τις καταχρηστικές πωλήσει. Ελπίζουμε ότι η ακρόαση θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ευχαριστώ όλους.